Dear uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τη δημόσια κρόση και πριν καλωσορίσω τους συγκεκριμένου επισκέπτες, έχω κάποια ανακοίνωση που ξέμεινα από χτες. Αφορά ερώτηση προς απάντηση για ποινική δίωξη κατά του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, 27 Οκτωβρίου, 12 μέλη υπέβαλαν γραπτή ερώτηση επευθυνόμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, σύμφωνα με τους κανόνες και απάντηση στην ερώτηση θα έπρεπε κανονικά να υποβληθεί εντός 6 εβδομάδων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται σήμερα αλλά αν η απάντηση δεν καταφθάσει να επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 130 σημείο 5, παράγραφος 5 του εσωτερικού κανονισμού και κατόπιν αιτήματος διαφόρων ομάδων, το θέμα θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο μερίσιας διάταξης της νέας ε, συνεδρίας, της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής. Θα δούμε όμως αν θα καταφτάσει σήμερα η ερώτηση και θα τροποποιηθεί η προσέγγιση αναλόγως, σας ενημερώσω εγώ. Πάμε στο σημείο 5 της διάταξης. Καλώς ορίζω του συγκεκριμένου φιλοξενούμενου μα στη δημόσια ακρόαση για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Χρηματοπιστωτική Εποπτεία. Αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σκοπό ακράσεω, η λήψη πληροφοριών από εμπλεκόμενου φορεί και εμπειρογνώμονε για τι συνέπειε τη πρακτική των προτινόμενων αλλαγών του Ευρωπαϊκού Συστήματο Χρηματοπιστωτική Εποπτεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας δίδει μεγάλη σημασία στο ζήτημα αυτό. Έχουμε δύο επιφανείς συνεισηγητές οι οποίοι εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της θητείας διότι έτσι θα δημιουργηθεί ένας βασικός πυλώνας για την ενίσχυση του υποπτικού συστήματος για το πρόγραμμα της ενιαίας κεφαλαγοράς και θα έχουμε αποτελεσματικότερο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας ούτως ώστε να προωθηθεί η χρηματοστική ολοκλήρωση και αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως αυτά που προέρχονται από το Brexit. Για αυτό το σκοπό Χαιρόμεθα ιδιαίτερος που φιλοξενούμε κάποιους επιφανείς επαΐοντες τον δόκτορα Ρίντι Καρδέιλ, καθηγητή για τις κεφαλογορές και τη σχετική νομοθεσία στο Λούντβικ Μαξιμίλιαν Πανεπιστήμιο του Μονάχου, πρόεδρος της ομάδας εμπλεκομένων φορέων ΕΣΜΑ, Σεμπαστιάν Αλμπέλα, πρόεδρος της Ισπανικής Επιτροπής για την αγορά των αξιογράφων, φιλή διευθύντρια του Finance Watch, Φέλιξ Χούφελτ, πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Μπάφιν και και ο Ζακ Ντελαζιέρ, εξίσου σημαντικός βεβαίως, παρόλο που είναι τελευταίος, πρόεδρος της ομάδας του Λιουπιπέδου του 2009 για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε μακροσκελή κατάλογο άλλων θέσεων που κατήχε. Είναι ιδρύτα, από τους ιδρυτές του ΕΖΑΣ και όχι μόνο αυτό. Τιμή μας που παρευρίσκεστε. Θα ξεκινήσουμε με παρουσιάσεις από τους φιλοξενωμένους και μετά θα δώσω το λόγο στους συνεισηγητές Περές και Μπάλσον. Ο δόκτωρ Ρούντιγκερ Βέιλ πρώτος έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά, ε. Επίτε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να συμμετάσχω στο πάνελ, για να συζητήσουμε την αναθεώρηση του ΙΖΑ, να δεχτούμε ότι ήταν ο κρογονιός λήθος της ευρωπαϊκής Συνομοθεσίας του Κοινοβουλίου αγορά, το ΙΣΑΣ, ε, πολύ σημαντικό επιτεύγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προτείνει αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχιτεκτονικής. Συμφωνώ ότι το Brexit και οι τεχνολογικές πρόοδοι και η προστασία των καταναλωτών και οι γενικοί στόχοι βιωσιμότητας θέτουν νέες ρυθμιστικές προκλήσεις. Και τώρα είναι και η ώρα να εξετάσουμε κάποια προβλήματα της διακυβερνήσεως του τομέα και πιστεύουμε ότι κάποιες από τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πηγαίνουν πολύ μακριά. Θα ξεκινήσω με την εξή πρόταση. Η ρυθμιστική υποπτήρα της ΕΣΜΑ να επεκταθεί σε νέους τομείς, θα έλεγα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει διάφορα επιχειρήματα που προβάλλει. Προβάλλει την οικονομική σημασία που έχει η βαθμολόγηση, εποπτική διατησία, κυρίως σε διασυνοριακές ε, περιπτώσεις, και ότι υπάρχει ανάγκη για πιο συνεπή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτά τα επιχειρήματα έχουν κάποια βάση, αλλά δεν είναι απόλυτα πιστικά. Το ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλύπτει πόρους και ταμεία, δεν δικαιολογεί ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κεντρική διαδικασία έγκρισης κάποιων προσφορών, κάποιων προϊόντων. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι καλύτερη η ευρωπαϊκή εποπτεία από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Διότι η σύνταξη ενό εγχειριδίου ε, είναι κάτι που σχετίζεται με το εθνικό δίκαιο. Οποιοδήποτε κίνδυνο που ε, απορρέει από εποπτική διατησία είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται από μέσα σύγκληση και να μην υπάρχει άμεση εποπτεία την ΕΣΜΑ. Από την άλλη, βέβαια, υποστηρίζω την πρόταση η εποπτεία τη ΕΣΜΑ επεκταθεί σε κρίσιμη βαθμολόγηση και θα πρέπει ΕΣΜΑ να είναι η μόνη αρχή αδειοδότηση και εποπτείας για υπηρεσίες ε, χορηγήσεως δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες ε, καλύπτουν όλη την Ευρώπη και έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οπότε έρχομαι στο επόμενο σημείο. Εποπτική σύγκληση. Στο μέλλον η πρόθεση εποπτικής σύγκλησης θα είναι βασικό καθήκον των ΕΙΣΑΣ. Βλέποντας την εξέταση των αποπλευράς που διεξάγει η ΕΣΜΑ, είναι προφανές πόσο σημαντικός είναι αυτός ο στόχος οι εθνικές πρακτικές διαφέρουν κατά πολύ συχνά και οι εκθέσεις της ΕΣΜΑ δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεως συμμορφώσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά έχει σαν στόχο τη βελτίωση των μέσων εποπτικής συγκλήσεως. Η νέα στατηγική εποπτική προσέγγιση διασμός είναι κάτι ε, φιλόδοξο και πολύτιμο. Βασικό πρόβλημα ποιο είναι, ότι το μέσο έχει σχεδιαστεί σε ένα είδος κολυσιεργίας που εμποδίζει την ταχεία κίνηση και τους εθνικούς φορείς να κινηθούν κατάλληλα. Είναι σαφές γιατί η Επιτροπή επιφορτισμένη με τις αναθεωρήσεις θα, είναι, θα αποτελείται αποκλειστικά προσωπικό της ΕΙΖΑ. Η προτινόμενη αλλαγή από εξέταση ομοτήμων προς ανεξάρτητη εξέταση δεν λαμβάνει υπόψη το ότι οι εθνικοί φορείς ελέγχου έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία όσον αφορά τις πρακτικές των αγορών, κάτι που είναι σημαντικό για τη διεξαγωγή αυτών των εκθέσεων και των ελέγχων. Τρίτο και τελικό σημείο της ομιλίας μου, η διακυβέρνηση των ε, φορέων αυτών. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διακυβέρνηση των ΑΕΖΑ να γίνει αποτελεσματικότερη, μετακινούμενη από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο λήψεω αποφάσεων στον τομέα εποπτική συγκλήσεω. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρέχει κάποια στοιχεία σύμφωνα με τον οποία αυτοί οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών προωθούν τα δικά του συμφέροντα ει βάρο τη ενώσεω κατά παρελθόν. Επίση, καθορισμό των καθηκόντων θέσπιση κανόνων και υποπτική συγκλήσεω σε δύο διαφορετικά μέρη ανεξάρτητα το ένα από το άλλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα. Υποστηρίζω ένθερμα ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου ΕΙΖΑ, αύξηση τη λογοδοσία στο επίπεδο 3 θεσπίσεως κανόνων και θέλουμε και εποπτικές εξουσίες να ανατίθενται στο εκτελεστικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο. Άλλος βασικός στόχος η βελτίωση συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων. Σημαντικότερο, θα πρέπει να διευκολύνουμε το κοινό έργο των ομάδων ενδιαφερομένων σε διατομιακά ζητήματα. Θα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και έγκαιρη συμμετοχή των ομάδων ενδιαφερομένων κύκλων στη διαμόρφωση κανόνων σε επίπεδα 2 και 3. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας το ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνει θεμελιώδη μετακίνηση από συντονισμό μεταξύ εθνικών φορέων υπό την αιγίδα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας προς εποπτεία των εθνικών αρχών από Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Τέτοιο τεράστιο βήμα προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιογράφων είναι κάτι πολύ πρόημο κατά την άποψή μου. Εγώ είμαι υπέρ εξελικτικής προσεγγίσεως προς επέκταση των εξουσιών του ΕΙΣΑ Ιδεοδός θα έπρεπε να προσέγγιση που εδράζεται επί καλά σχεδιασμένων, συνεκτικών και καλά εξετασμένων, εξεταστησών μάλλον εθνικών ε, στρατηγικών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σεμπασιάν Αλμπέλα, ο πρόεδρος της Ισπανικής Επιτροπής Αγοράς Κινητών Αξιών. Έχετε το λόγο. το μικροφόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι τιμή για μένα που απευθύνομαι προ εσά ω πρόεδρο τη Ισπανική Επιτροπή Αγορά και των Αξιών CMNV και εκτιμώ την ευκαιρία που μου δίνεται να συμμετέχω στην ε, πρόταση, στη συζήτηση τη Επιτροπή σα για την πρόταση μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Χρηματοοικονομική ε, Εποπτεία. Να σα πω πώ θεωρούμε, και ποια είναι η υπόψη μα για τη μεταρρύθμιση. Να σα πω ότι υποστηρίξουμε το project τη ενιαία χρηματοοικονομική αγορά και το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και Θέλουμε προφανώ και εμεί να ενισχυθεί η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, οτιδήποτε έχει ως σκοπό να κάνει την ΕΣΜΑ πιο ευέλικτη και πιο δυνατή, πιο ισχυρή στον συντονισμό των εθνικών ευρωπαϊκών αρχών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθεί αυτό, αυτή η τελεστική επιτροπή η οποία θα αποτελέσει το κινητήριο μηχανισμό αν θέλετε πίσω από την ενίσχυση. Το η Επιτροπή των Εποπτών θα πρέπει να παραμείνει το πιο υψηλό βαθμό όργανο για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΣΜΑ. Ωστόσο καταλαβαίνουμε και υποστηρίζουμε τα νέα εργαλεία τα οποία ε, παρουσιάζονται στην πρόταση για την ενίσχυση και τη συντονισμό των ε, ρόλων για την πρόθεση της σύγκλησης της ΕΣΜΑ και αποδεχόμαστε την αλλαγή της προσέγγισης από ένα σύστημα αξιολόγησης αμοτήμων σε ένα σύστημα το οποίο θα ηγείται η ΕΣΜΑ. Επίσης, συμφωνούμε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να εγκρίνει με την συμμετοχή της Επιτροπής των Εποπτών τα στρατηγικά σχέδια για να αποτελέσουν αυτά το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν οι εθνικές αρχές, αρκεί οι εθνικές αρχές να μπορούν να προσθέσουν προφανώς και προτεραιότητες και στόχους. Επίσης πιστεύουμε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο ενεργά τα εργαλεία όπως η παραβίαση του κοινωτικού δικαίου και τη σχετική απόφαση η οποία θα ανταποκρίνεται στη λειτουργία της Εκκληστικής Επιτροπής. Άρα, όντως, η ΕΣΜΑ θα πρέπει να συμμετέχει πιο πολύ στην εποπτεία των CCPs και να αναλάβει νέε ευθύνε άμεση εποπτεία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη σχέση με τρίτε χώρε, σε ό,τι αφορά του κρίσιμα ορόσημα κτλ. Ωστόσο, υπάρχουν δύο τομεί όπου δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ούτε ανάγκη ούτε όφελο αν γίνει αυτό. Μιλάμε για κάποια είδη αξιών και σε ό,τι αφορά τα προσπέκτουσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διάφορα εργαλεία για επιχειρηματικά κεφάλαια και για επενδυτικά κεφάλαια, UVECA, USEF, LTIF. Αλλά δεν βλέπουμε το λόγο μόνο και μόνο επειδή θεωρούνται ευρωπαϊκά και ρυθμίζονται άμεσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι το παραδοσιακό σύστημα που βασίζεται στην αμοιβή αναγνώριση αρκεί. Και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τέτοια διάκριση σε ό,τι αφορά την εποπτεία των ε, διευθυντικών εταιριών και προϊόντων. Ο δεύτερος τομέας, τα προσπέκτους, ε, μια προτάση η οποία δεν αναφέρθηκε στην προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος να υπάρξει να αναλυφθούν αυτά τα καθήκοντα από την ε, ΕΣΜΑ. οι εθνικές αρχές, όπως η Ισπανική για παράδειγμα Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών, έχουν την εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Οι εθνικές αρχές λοιπόν γνωρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ποιοι είναι οι εκδότες, και ποιο είναι και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα εγκρίνει τους ε, εγκεκριμένους, εξειδικευμένους εκδότες που περιλαμβάνει και, για παράδειγμα, τις εταιρείες ε, και πιστεύουμε ότι το θέμα των προσπέκτους έχει να κάνει και με την οικονομική κατάσταση των εκδοτών. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τονίζει την ανάγκη ενοποίησης του συστήματος για να υπάρξει μια πραγματική αγορά, ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά, ενιαία κεφαλαία αγορά. Συμφωνώ αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα θα πρέπει να δημορφωθούν σε ένα κεντρικό επίπεδο. Και μόλις λοιπόν ε, συμφωνήσουμε για την πορεία και για τους στόχους, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να σεβαστεί και τον εποπτικό ρόλο του σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν στεναρά εποπτικά όργανα με τις ε, αντίστοιχες αρμοδιότητες προκειμένου στην Ευρώπη να συνεχίσουμε να έχουμε μια ποικιλομορφία αγορών και οικονομικών κέντρων. Αυτό είναι πολύ κεντρική σημασία αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή κεφάλαια αγορά με μεγαλύτερη διείσδυση, η οποία πραγματικά θα συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων, όχι μόνο στην πρόθεση των μεγάλων εταιριών. Και να περιοριστεί το επίπεδο εξάρτηση από τη χρηματοδότηση από τους τραπεζών Σα Ευχαριστώ και φυσικά είμαι στη διάθεσή σα αν θα έχετε ερωτήσει. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ομιλία την κυρία Αμφιλή από την Finance Watch. Η Final Watch καλωσορίζει τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε αυτή την ε, ακρόαση. Πιστεύουν ότι ο του Ευρωπαϊκού Συστήματο Χρηματοοικονομική Εποπτεία είναι σημαντική πρωτοβουλία υπό το φω ε, των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα με τη δημιουργία των ΑΕΖΑΣ. Από το σκοπό του δημοσιονομικού κανονισμού και τη εποπτεία είναι να εξασφαλίσουμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, εκεί όπου οι καταναλωτέ, οι επενδυτέ και οι φορολογούμενοι ε, θα πρέπει να προστατεύονται παρκώς. Για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη του στόχου χρειαζόμαστε ισχυρέ ευρωπαϊκέ αρχέ, οι οποίε έχουν καλή στελέχωση και χρηματοδότηση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε κάποια απογοήτευση, ελλείψη φιλοδοξία που παρουσιάζεται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη πριν την υποβολή της προτάσεως εμπεριέχει συστάσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει αλλαγή αλλά η πρόταση τελικά δεν είναι τόσο φιλόδοξη όσο ήταν αρχικά. Θα θέλαμε να δούμε αναζωγόνηση της ομάδας υψηλού επίπεδου χρηματοοικονομικής εποπτείας. Αυτό θα επέτρεπε στους ειδικού να σκεφτούν ποιες εξελίξεις είχαμε από την αρχική έκθεση μέχρι τώρα και να κάνουν συστάσεις για βελτιώσεις. Υπάρχουν αρκετοί τομείς που η Financial Watch ε, πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν βελτιώσεις. Καταρχάς, Πιστεύουμε ότι ο ενεργός ρόλο των Αιζα και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βοήθησαν την εναρμόνιση ε, της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Όμως παραμένει ένα κενό όσον αφορά την εποπτεία αυτή. Ο καθορισμός άλλων συστημικών θεσμών που είναι σημαντική παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρμοδίων αρχών. Παρά τι κατευθυντήρε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα υπάρχουν διαφορέ όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων, όσον αφορά τη συστημική σημασία που έχουν οι διάφοροι φορεί. Αυτό επηρέασε επίση και τι αρχέ των κρατών μελών, διότι χρησιμοποιούν τα CDR και το CRR ε, και ε, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στα διάφορα κράτη. Χρειάζεται αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εναρμονισμένη προσέγγιση, κάτι περισσότερο από τώρα. Γι' αυτό θα θέλαμε να δούμε ισχυρότερο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, Συστημικού Κινδύνου. Θα πρέπει οι εθνικοί φορείς να παίζουν πιο ενεργό ρόλο στον εντοπισμό των συστημικών, ε, συστημικά σημαντικών θεσμών και να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία, τα μακροοικονομικά. Και μετά η Financial Watch μαζί με ΜΚΟ που εκπροσωπούν τους καταναλωτές θα ήθελε να δει μεγαλύτερο ρόλο για τους ΕΙΖΑ στην πρόθεση προστασίας των καταναλωτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φορεί αυτοί, οι ΕΙΖΑ, θα πρέπει να προωθήσουν σύγκληση εποπτική όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικότητα ώστε όλες, όλοι οι χρήστε χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να αντιμετωπίζονται δίκαια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη δεσμευτικών τεχνικών προδιαγραφών για την ε, λειτουργία των επιχειρήσεων και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό βάσει των προτύπων. Πιστεύουμε επίση ότι οι ΑΕΖΑ θα πρέπει να έχουν ε, τη δυνατότητα να απαγορεύσουν, να περιορίσουν χρηματοπιστωτικέ δραστηριότητε που είναι ει βάρο των καταναλωτών. Ισχυρότερη εντολή για προστασία των καταναλωτών προποθέτει επίση διαθροτικέ μεταρρυθμίσει. Προτείνουμε λοιπόν κάθε δικημβούλιο ίσας να καταρτίζει μόνιμη επιτροπή που θα παρτίζεται από εθνικές αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνε για την επιβολή των αρχών προστασίας καταναλωτών. Για να εξασφαλίσουμε το ότι η προστασία των καταναλωτών τελικά θα επιτυγχάνεται, οι ΕΖΑΣ θα πρέπει να δίνουν τους αναγκαίους πόρους θα διαθέτουν αναγκαίου πόρου. Το 20% τουλάχιστον των προπολογισμών των αρχών θα πρέπει να διατίθεται για την προστασία των καταναλωτών. Η Finance Watch πιστεύει ότι οι ASAS θα πρέπει να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην πρόθεση βιώσιμης χρηματοδότησης, χρηματοπιστωτικών ε, ενεργειών, λαμβάνοντα υπόψη παράγοντες διακυβέρνηση και κοινωνικούς στόχους ευρύτερους. Θα θέλαμε οι ASAS να παρακολουθούν τάσεις που διαπιστώνονται στους διάφορους τομείς. Εν τέλει, όσον αφορά τη συμμετοχή των κύκλων ενδιαφερομένων και τη συμμετοχή του στις ASAS, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις ομάδες που εκπροσωπούν τους εμπλεκομένους να εξετάζουν τις ε, κανόνες που θεσπίζουν οι ίσας. Θα πρέ... Δεν θα πρέπει όμως τελικά οι κύκλοι των ε, εμπλεκομένων φορέων συμμετέχουν τόσο πολύ στη διαμόρφωση των κανόνων. Χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση. Θα πρέπει καταναλωτές και το των, ε, και εκπρόσωποι των διαφορετικών κύκλων συμμετέχουν και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στους, ε, στις ομάδες αυτές των κύκλων των ενδιαφερομένων. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Χούφελτ, ο πρόεδρος της Παθήν. Πρόεδρε, βουλευτέ, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ ιδιαίτερα που με καλέσατε σήμερα για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα το θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ευρωπαϊκής Υποπτείας, Χρηματοοικονομικής Υποπτείας. Και είναι μεγάλη τιμή μου που το κάνω αυτό μαζί με τον αρχιτέκτονά του συστήματος, τον Ζοκ Ντελαροζιέρα. Και μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά το οικοδόμημα των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών, των ΕΣΑ. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι πολλοί από του συναδέλφου μου στη ΠΑΦΗΝ και εγώ ίδιο, είμαστε πολύ παθιασμένη, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοοικονομική εποπτεία και τον, ε, χρηματοοικονομικό κανονισμό στην Ευρώπη και γενικότερα, καθώς και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Θέλουμε να σταθούμε επιτυχία. Θεωρούμε ότι αφαιρώνουμε ένα σημαντικό τμήμα της ενέργειάς μας και του χρόνου μας για να βελτιώσουμε την, το εγχείρημα αυτό. Προφανώς ε, εκπροσωπώ μια μεγάλη εθνική αρχή, αλλά δεν θα ήθελα στις παρατηρήσεις μου να θεωρήσω ότι είμαι εγώ, εμείς ε, κατά ημών, ε, ότι αποδιόμαστε σε ένα πόλεμο εθνικών εναντί ευρωπαϊκών συμφερόντων. Αλλά θα ήθελα να σας προσεγγίσω πέντε αρχές σε ό,τι αφορά την οτροπία μας για τη λειτουργία των ε, Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών. Καταρχά, μην προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να φτιάξουμε κάτι το οποίο λειτουργεί. Δεν μπορώ να επιβεβαίωσω ότι συστηματική παραβίαση υπάρχει και υπέρβαση των αρμοδιατήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όπως υπονοούν κάποιοι. Αλλά δεν πιστεύω να πω ότι υπάρχει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη αρμοδιοτήτων ε, και τα δύο θεωρώ ότι είναι υπερβολικά. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις αρμοδιότητες που ήδη έχουν, όχι συστηματικά να διευρύνουμε το πεδίο των αρμοδιότητων τους. Κατά δεύτερον, να μην υπάρχει επόπτης του επόπτη, ο εποπτεύων του υποπτεύοντος. Όποιος θέλει να δημιουργήσει επόπτης ε, των εποπτεύοντων, ουσιαστικά ε, υπερβάλλει, οι διαδικασίες, οι δομές και ο σχεδιασμός, όλα αυτά προαπαιτούν κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες όμως ε, στην πορεία θα απαλείψουν ε, τη φύση, τον, τον ρόλο των ε, μέλων της ΕΖΑ. Και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε για να μην υπάρχει μια σύμμετρη προσέγγιση. Κατά τρίτο να μην υπάρχει ε, το γραφειοκρατικό τέρας, γιατί η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, οι πολύ περίπλοκες διεπαφές σε βασικές διαδικασίες εποπτείας, όπως ε, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η εσωτερική έγκριση μοντέλων, το outsourcing, θα δημιουργούσαν τεράστιες ανεπάρκειες, κόστος, γραφειοκρατικό άχθος και καθυστέρηση. Πολύ απλά θα πρέπει να μην στραφούμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Κατά τέταρτον, ρύθμιση έναντι Θα πρέπει να σεβαστούμε την ακαιρεότητα του κανονιστικού πλαισίου έναντι της εποπτείας και αντιστρόφως, αλλά να μην τα μπλέξουμε, γιατί αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Η σχέση μεταξύ έκτα ως επόπτη και είπα ως ρυθμιστή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και συνέχεια το υπενθυμίζω αυτό στους συναδέλφους του, της Υποπτικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Αλλά αυτό έχει συνεπείς και στη χρηματοδότηση, γιατί η εποπτεία ουσιαστικά χρηματοδοτείται από εισφορές των ε, σχετικών ε, θεσμικών οργάνων, ενώ ε, η ρύθμιση ουσιαστικά προέρχεται από τα χρήματα του φορολογουμένου. Να μην τα μπλέκουμε αυτά κατά πέμπτον. Να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ όπου υπάρχει διαφορετικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν παραδείγματα όπου ο ρόλο των ε, εσά, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, λόγω τη ευρωπαϊκή του ε, φύση, θα έπρεπε να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αντιστοιχία τρίτων χωρών. Η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, για τρίτες ε, χώρες όπως σε χρηματοοικονομική ανάλυση δεδομένων. Θα πρέπει να ενισχυθεί επίσης ανάπτυξη μιας κοινή χρηματοοικονομικής ε, γλώσσας. Αυτό χρειάζεται όχι μόνο στα πλαίσια της ΕΣΜΑ, αλλά γενικότερα. Άρα ουσιαστικά να πούμε ότι απορρίπτουμε οποιαδήποτε απόπειρα να προσθεθεί κόστος, περιπλοκή, άχθος και θεωρούμε ότι τα μέλη μάλλον η προσέγγιση της, ε, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών βάσει των μελών της αποτελεί ένα απαραίτητο πύλωνα και υποστηρίζουμε την ενίσχυση του ρόλου, του ρόλου των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα ο κύριος Ντελαροζιέρα έχει το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές έχουν διδραματίσει σημαντικό ρόλο πρόθεσαν τη δημιουργία και την υλοποίηση κοινών κανόνων για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ευρέω ε, αναγνωρισμένο. Θα ήθελα λοιπόν ότι ίσως θα έπρεπε σαφέστερα από ό,τι στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να εντοπίσουμε εμείς τους στόχους και τους ρόλους των διαφόρων εποπτικών αρχών. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή, η ΕΜΠΑ λοιπόν κάνει τη δουλειά της Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών κάνει ό,τι μπορεί, ίσως όχι αρκετά, όσον αφορά την εποπτεία και τη σύγκληση την εποπτική. Για την ΕΟΠΑ, την βλέπω αυτή κάπως σαν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θα πρέπει να εστιάζεται επί κοινών ορισμών και ερμηνείας προτύπων, και εναρμόνιση ρυθμιστικών απαιτήσεων. Αλλά διστάζω επί μιας προτάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καθιστά την ΕΙΟΠΑ εκείνο τον φορέα που εγκρίνει εσωτερικά πρότυπα και μοντέλα. Θα ήταν εσφαλμένο αυτό, διότι η αξιολόγηση εσωτερικών μοντέλων και η έγκρισή τους από την ΕΙΟΠΑ θα κατακαιρματίζεται και θα απομονώνεται από την καθημερινή εποπτεία των εθνικών αρχών ελέγχου και κάτι τέτοιο θα δημιουργεί κάποια αναποτελεσματικότητα. Όσον αφορά την ΕΣΜΑ, η κατάσταση διαφέρει κάπως, διότι πέρα από τον καθορισμό προτύπων και από την εποπτική σύγκληση, υπάρχει περισσότερο περιθώριο για άμεσα εποπτικά καθήκοντα, δοθήσεις της διασυνοριακής διαστάσεως ε, πολλών δραστηριοτήτων των κεφαλαγορών και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη κοινού εποπτικού φορέα, όπως το SSM. Κατά την άποψή μου λοιπόν, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε βελτιώσεις, οι οποίες βελτιώσεις ίσως υποστηρίξουν την εφαρμογή ενιαίων χειριδίου κανόνων και αντίστοιχες ρυθμίσεις με τρίτες χώρες. Αν δείτε λοιπόν τις ε, προτάσεις από αυτή την οπτική γωνία, εγώ θα έλεγα ότι ναι, είναι καλό ε, να αυξηθεί η ιδιαιτησία, η λήψη αποφάσεων, οι ερευνητικές εξουσίες που θα έχουν οι εποπτικές αρχές σε κάποιους τομείς, όπως είναι οι παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, διευθέτηση διασυνοριακών διαφωνιών, και συνεπής εφαρμογή των προϋποθέσεων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικότατο σημείο. Μου είπαν ότι κάποιοι από τους ούτως αποκαλούμενους κοινού κανόνες που θεσπίζονται από τις αρχές δεν ακολουθούνται από τις εθνικές αρχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Δεν είμαι σίγουρος αν μια θεμελιώδης με αλλαγή των διοικητικών δομών ε, διαχείρισης των, εθνικών, των υποπτικών αρχών είναι κάτι καλό και το να δημιουργήσουμε νέο φορέα που θα προσθέσει μια ακόμη στιβάδα στο σύστημα ε, και θα περιπλέκει το όλο σύστημα ότι είναι κάτι καλό. Θα πρότεινα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, να αυξηθεί η ανεξαρτησία του φυσταμένου Διοικητικού Συμβουλίου με μια προσθήκη, Φερρυπίν, δύο ή τριών ανεξαρτήτων μελών που θα προέρχονται από ανεπιστημιακούς και επιχειρηματικούς ε, κύκλους. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα καλό όχι για την θέσπιση κανόνων, διότι αυτό πραγματικά βρίσκεται στα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά για την αποσύνδεση και την εξομάλυνση διαφορών ε, ε, ερμηνείας και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Η προσθήκη δύο ή τριών μελών έξωθεν με μεγάλη ανεξαρτησία θα προσέθεται μια διάσταση ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας. Τέλος, νομίζω ότι η ιδέα του να δοθούν άμεσες εποπτικές εξουσίες σε διασυνοριακές ε, δραστηριότητες όπου υπάρχουν συνέργειες σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ξέρω αν είναι καλό η αύξηση των εξουσιών εποπτείας των ευρωπαϊκών φορέων εποπτικών και κυρίως της ΕΣΜΑ έχει νόημα εκεί που η ευρωπαϊκή προσέγγιση δίνει πραγματική προστιθέμενη αξία. Συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κάποιοι άλλοι φορείς όπως οι πάροχοι δεδομένων, οι διαχειριστές συστημάτων βαθμολόγησης θα μπορούν να εποπτεύονται άμεσα από την ΕΣΜΑ δοθέντων των προναφερθέντων κριτηρίων. Αυτό ισχύει και για κάποιες υποδομές χρηματιστηριακών αγορών που έχουν μια έντονη συστημική και διασυνοριακή διάσταση, όπως τα CCPs που θα ελέγχονται καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω την πρόταση που έγινε πρόσφατα, ούτως ώστε η ΕΣΜΑ να παίζει έναν άμεσο ρόλο όσον αφορά την εποπτεία των διασυνοριακών CCP της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των χωρών με την υποστήριξη βεβαίως κεντρικών τραπεζών που είναι σημαντικό. Επίσης, όπως και κάποιοι από τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως, Είμαι διστακτικός όσον αφορά την επέκταση της άμεσης εποπτείας από την ΕΣΜΑ και σε άλλους τομείς, όπως είναι αδειοδότηση κάποιων κατηγοριών ταμείων ή ε, κάποιων εγχειριδίων και φυλαδίων. Ε, αυτό ίσως να οδηγεί σε αντιθέσεις και ανεπάρκειες και προβλήματα μεταξύ των ε, αρμοδίων εποπτικών φορέων. Τρία σημεία στο τέλος. Το πρώτο, δημοσιονομικές συνέπειες. Συμφωνώ με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, 60% του προπολογισμού να πηγαίνει ε, στον τομέα της, ε, το βιομηχανικό και στον έλεγχο αυτού του τομέα. Δημοσιονομική εποπτεία θα πρέπει να διενεργείται από τους εθνικούς φορείς ελέγχου. ESRB, το σημείο θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του ESRB έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως μέσω διορισμού επιφανών εμπειρογνωμόνων και δεν θα πρέπει περαιτέρω να ενταχθεί στη λειτουργία της ΕΚΤ το ESRB που προτείνεται. Θα είναι λάθος κάτι τέτοιο. Και τέλος, κατεπίγουση ανάγκη η θεσπίσεως μέτρων αυτών που συζητούμε σήμερα, ούτω ώστε να αναθεωρηθεί η λειτουργία των εθνικών υποπτικών αρχών, ε, των ευρωπαϊκών υποπτικών αρχών. Αυτή η πρόταση πρέπει να υιοθετηθεί στα πλαίσια της θητείας της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και όντως ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στην νομοθετική διαδικασία πιστεύω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό πριν το τέλος της θητείας και σε αυτό έχουμε αποφασίσει και γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές για το μεγάλο εύρος των παρατηρήσεών τους μας ε, παρουσίασαν και διαφορετικές προοπτικές, αλλά είχαν και κοινά στοιχεία στις ε, παρεμβάσεις τους. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση μαζί σας και ασφαλώς ε, συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια που έγιναν, αλλά θα πρέπει να δούμε τι είναι εθνικό, τι είναι διευρωπαϊκό, για να μην υπάρχει στατική προσέγγιση. Θέλουμε πιο πολύ διασυνοριακή ενσωμάτωση των κεφαλαίων αλλά προφανώς ε, η επικουρικότητα, η αναλογικότητα και όλα αυτά είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το έργο μας και ασφαλώς και ισχύουν και εδώ στον τομέα αυτό. Οι μας τώρα. Ο κύριος Μπάλτς, καταρχάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα ως εισηγητής ε, του ΕΛΚ και με την συνεισηγήτρια την κυρία Περές να σας καλωσορίσω εδώ στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Τότε στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής ήμουνα ήδη από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέλος της διαπραγματευτική ομάδας και η εντύπωση που είχε αφήσει τότε η χρηματοοικονομική κρίση είχε ω αποτέλεσμα καταρχάς τον, τον οργανισμό για τι Ευρωπαϊκέ Επιλεκτικές Αρχέ το 2010, μία από τις πρώτες αντιδράσεις. από τότε έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και η συγκυρία στην Ευρώπη και η πολυπλοκότητα έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα πρέπει και το οικοδόμημα της εποπτείας να εξεταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από το διεθνές επίπεδο για τα μεγάλα ιδρύματα θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στο εθνικό επίπεδο βασικά. Και θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί το εξής. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές και ο ρόλος των δύο πλευρών να παραμείνει σε συνάρτηση και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των προτύπων, θα πρέπει να δούμε και τις προτεραιότητές μας Μήπως ε, θα πρέπει να αστιαστούμε πιο πολύ στην ε, υλοποίηση των υφιστάμενων ε, κανονισμών. Αυτή λοιπόν η μεταρρύθμιση αποτελεί μια ευκαιρία για τη διευκρίνηση και των μελλοντικών αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών και από πλευρά του συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι εκπροσωπώ πολλού συναδέλφου λέγοντα αυτό. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα των ε, αρχών αυτών. Να σας ευχαριστήσω όλους σας που ήλθατε εδώ σήμερα για να μοιραστείτε μαζί με μας ε, την εμπειρογνωμοσύνη σας, την εμπειρία σας κυρίως. Και γι' αυτό λοιπόν οι ερωτήσεις μου θα επιδοθούν κυρίως σε τρία σημεία. Πρόεδρε, ως συνεισηγητής, αν θα μου επιτρέπετε, επιτρέψετε να μιλήσω λίγο παραπάνω. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον κύριο Ντελαροζιέρ σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξετε. Είναι το εξή. Κυρίω θα πρέπει να κοιτάξουμε την ε, διακυβέρνηση, την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Πέρα από το, ε, την Επιτροπή Εποπτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και μια εκτελεστική επιτροπή. Το ένα να είναι υπεύθυνο για τα θέματα ρύθμιση και το άλλο να είναι θέματα υπεύθυνο για θέματα εποπτείας. Αλλά λείπουν οι μηχανισμοί ελέγχου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Πώς λοιπόν κύριε Ντελαροζιέρ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον θα υπάρχει καλή διακυβέρνηση στους οργανισμούς αυτούς. Προς τον καθηγητή Βάιλ τώρα. Να θέσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ε, λέει ότι αυτή η πρόταση αποτελεί, για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους αποτελεί την ε, πρόταση της και τη συμβολή της για την εναλλαγικότητα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής αξίωση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των κανονισμών. Πώς λοιπόν μπορεί να υπάρχει αναλογικότητα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τις ε, διευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αναλογικότητα σε ό,τι αφορά και την ε, λειτουργία των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών προ τον κύριο Αλμπέλ. Να ρωτήσω το εξή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ το συντονισμό των εθνικών αρχών με τις Ευρωπαϊκές Υποπτικές Αρχές χωρίς ε, ε, σαφή ρόλο των εθνικών ε, υπηρεσιών ούτε στο μέλλον θα μπορέσουμε να λειτουργούμε όπω και τώρα. Πώ λοιπόν θα αποφύγουμε την αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων, πώς θα την περιορίσουμε και τέλος, τελευταίο ζήτημα προς την κυρία Φιλή. Προηγουμένως στην εισήγησή σας μας είπατε ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν καλύτερη χρηματοδότηση και πιο πολύ προσωπικό. Πείτε μας λίγα παραπάνω για το θέμα αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, οι αντισυμβαλών, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει ε, να βελτιωθούν. Πείτε μας, κάντε μας μερικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Περέζα. Merci, merci beaucoup de vos contributions, euh, chers euh, experts, chers... Euh. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας. Ε, μπαίνουμε στην καρδιά αυτής της μεταρρύθμισης που όπως πολύ πιστεύω και εγώ ότι, ε, ότι θα μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε πριν το τέλος αυτής της θητείας για πολλούς και διάφορους λόγους. Όχι μόνο για να έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας αλλά και επειδή Πρόκειται για μια πολύ αναμενόμενη μεταρρύθμιση η οποία συμβαδίζει με μια πιο μεγάλη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία στηρίζει το Κοινοβούλιο δηλαδή το να μπορέσουμε όχι μόνο να ολοκληρωθεί η Ένωση αλλά και να γίνει και μια πρώτη ε, έναρξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κεφαλαγοράς. Θυμάμαι όταν ε, η Κομισιόν ανακοίνωσε το πρώτο ε, πράσινο βιβλίο για την ένωση των κεφαλαγορών ε, ε, κανείς δεν είχε καν σκεφτεί αυτή την ιδέα και βλέπουμε πως σιγά σιγά ε, κομμάτι κομμάτι αυτές οι κεφαλαγορές ενώνονται και περί αυτού πρόκειται χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και το πλαίσιο του Brexit. Να προσθέσω ένα επιχείρημα που για μένα αποτελεί το νήμα που ενώνει ολόκληρη αυτή τη συζήτηση γιατί είναι το θέμα της σύγκλησης γιατί θα πρέπει να το να γνωρίσουμε μεταξύ μας το κόστος μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι τεράστιο. Αφιερώνουμε ώρες και ώρες για να ξεκινήσει μια πρόταση, για να εγκριθεί και στη συνέχεια για να εφαρμοστεί. Αλλά αφού έχουμε φτιάξει και έχουμε ανέβει το βουνό και ξαφνικά κατρακυλάμε και πάλι προς τα πίσω επειδή υπάρχει μεγάλη απόκληση στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, ε, τότε όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει εκμεδενίζεται. Γι' αυτό και το θέμα της σύγκλησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε. Έχω όμως την εντύπωση ότι το να δούμε πώς θα γίνει η σημερινή διακυβέρνηση ε, των ε, ε, οργανισμών, πώς μας οδηγεί στο να λειτουργήσουν όλα αυτά, δεν είναι η καλύτερη δυνατή και ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει τα πράγματα. Να προσθέσω κάτι ακόμα, μια ανησυχία που ίσως δεν ήταν προτεραιότητα όταν άρχισαν να λειτουργούν οι διάφοροι οργανισμοί, ότι δηλαδή σήμερα Έχουμε το θέμα της προστασίας των επενδυτών ή των καταναλωτών, όπως θέλουμε να τους πούμε. Όντως αυτή η διάσταση νομίζω ε, πρέπει να ε, ενδυναμωθεί. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ε, ανάπτυξη της καινοτομίας στην αγορά. Το fine tech όπως το λέμε τώρα. Και Επίσης το θέμα της βιώσιμης οικονομίας όπως την ονομάζουμε, πώς θα μπει στην εντολή των οργανισμών πέρα από την νομοθεσία αναφοράς. Τώρα, πιο ειδικέ ερωτήσεις. Κύριε Κυρβάλη, ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις σας. Εσείς υποδείξατε φιλικά στα συμπεράσματά σας ότι δεν θέλετε να περάσετε από συντονισμό σε εποπτεία των ε, εθνικών ελεγκτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως όμως για να βάλουμε, φτιάξουμε μια ενιαία, ενιαία κεφαλαγορά ακριβώς θα έπρεπε Αφού κάνουμε αυτή τη δύσκολη νομοθετική εργασία της εναρμόνισης, μήπως και η ενίσχυση της εποπτείας και η δυνατότητα ευρωπαϊκής εποπτείας ε, όσον αφορά τη σύγκληση αυτών των νομοθεσιών θα ήταν κάτι το σκόπεμο. Και ε, στη συνέχεια είπατε επίσης ότι δεν θέλετε τον ε, αρχιχωροφύλακα τον, τον επόπτη των εποπτών. Ναι, ωραία. Υπάρχει εξωσημείωτη πυρογνωμοσύνη, αναγνωρισμένη κτλ. Όμως πιστεύετε ότι το ίδιο ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές ε, εθνικές αρχές ελέγχου και εποπτείας. Πιστεύετε ότι ε, χωρίς να δικαταστήσουν τις εθνικές αρχές οι ευρωπαϊκές, μήπως αυτή η εργασία εποπτείας επαλήθευσης ε, της κατάστασης των μέσων των συνθήκων εφαρμόγης των ε, ευνίδιων ελέγχων και τα λοιπά θα μπορούσαν να γίνουν από αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή που θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε. Σεμπαστιάν Αλμπελά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτον, τι πιστεύετε για την ε, αρχιτεκτονική των διατάξεων για την εποπτεία των ΣΕΣΕΠΕ ε, και ιδιαίτερα MR2, ε, αυτά που προτείνονται μάλλον με το MR2, Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγχώνευση των δύο θέσεων και για παράδειγμα να προβλέψουμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως ε, υπεύθυνο για το ΣΣΠ. Τώρα, για τα σε εσεί δεν είστε ο μόνος που εκφράσατε δισταγμού σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν η εξή. Ε, όσον αφορά τα φυλάδια, ε, εγώ καταλαβαίνω ότι ναι, όταν είμαστε πιο κοντά στην αγορά καταλαβαίνουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Όμως δεν χρειάζεται πιστεύετε αυτό το ε, πνεύμα της σύγκλησης να αναπτυχθεί και για αυτά τα φυλάδια και τα βιβλία και αν, αποσύρουμε αυτή τη λογική της εποπτείας, ποιοι θα είναι οι όροι για να βελτιωθεί η σύγκληση. Έπειτα, μιλήσατε για το stakeholders group. Ποιο θα ήταν η σωστή συνεισφορά στην πρόταση της Κομισιόν, γιατί κατά με αυτό παραμένουν φέζονες. Ξέρω ότι δίνονται, κάποιες, δίνονται εδώ κάποιες αρμοδιότητες, αλλά ποιες θα πρέπει να είναι αυτές ακριβώς. Οι συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν που ίσως μπορείτε να υποβάλλετε θα ήταν ευπρόσδεκτες. Επίσης προτείνατε κάθε ε, υποπτική αρχή να, και η Επιτροπή της ε, που ασχολείται με τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι εθνικές δηλαδή αυτές οι ε, εποπτικές αρχές, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ενισχυμένος πόλος μέσα στην, ε, στη ΕΣΜΑ για να ενισχυθεί αυτή η λειτουργία. Φέλιξ Βελφέλτε δύο ερωτήσεις επίσης. εσείς είχατε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αρχή επόπτης. Ο επόπτης όλων των εποπτών. Άρα λοιπόν σε εσά ε, απευθύνεται αυτή η ερώτηση ε, που έκανα πριν, ότι δηλαδή δεν θα έπρεπε να, ε, να υπάρχει μια δυνατότητα επιπλέον ελέγχου εφόσον οι εθνικές αρχές δεν έχουν οικονομικά τις δυνατότητες. Λοιπόν, μιλήσατε τώρα για τη ρύθμιση. Σημαίνει αυτό ότι συμφωνείτε για τη χρηματοδότηση της ρύθμισης ε, των, ε, της εποπτείας από τις αρθενικές αρχές ε, ενώ θα πρέπει να συμβάλλουν οι φορείς της αγοράς στη χρηματοδότηση της εποπτείας. Έπειτα για το τραπεζικό συμβούλιο, ε, την τραπεζική αρχή, συγγνώμη, ε, έχετε προτάσεις συγκεκριμένες όσον αφορά την εντολή, γιατί το είδαμε χτες και στην ενταλλαγή απόψε με τον Μάριο Ντράγκη, θεωρούμε ότι έχουν μια λειτουργία επεξεργασίας πριν, αλλά που δεν λαμβάνονται ακριβώς υπόψη από τους φορείς της αγοράς. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Τέλος, για το ΣΣΠ, Σας θέτω την ίδια ερώτηση όπως στον προηγούμενο μιλητή. Θα συμφωνούσατε να ανατεθεί σε ένα μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου όπως θα έχει αναδιαρθρωθεί γύρω από το διοικητικό συμβούλιο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες όσον αφορά το ΣΣΠ. Thank you. Um, I think uh, we already received... Νομίζω Λέει ο Πρόεδρο ότι ε, ακούσαμε αρκετέ ερωτήσει, οπότε να έχουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων και μετά συνεχίσουμε με τους σκιώδει για έναν δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων προς τους ομιλητές μας, προς μα. μας. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, να αρχίσουμε πάλι με την ίδια σειρά. Παρακαλώ. Thank you very much uh, to the um, Ευχαριστώ πολύ τους συνεισηγητές. Πολύ σημαντικές οι ερωτήσεις τους και πολύ δύσκολες. Το θέμα της αναλογικότητας. Πώς εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη αναλογικότητα. Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές, οι συνομοθέτες ε, έχουν τον έλεγχο στα χέρια τους. Μπορούν στο πρώτο επίπεδο να καθορίσουν τα καθήκοντα για τους εποπτικούς φορείς να βάλουν λεπτομέρειες, να αναφέρουν τι πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 2 αλλά και σε επίπεδο 3. Αυτό συμβαίνει περιστασιακά όμως. Η πρώτη μου πρόταση θα ήταν αυτό να εξεταστεί περαιτέρω. Μήπως και άλλες συστάσεις και άλλοι προσανατολισμοί και ερωταπαντήσεις και κατάλογοι αν όλα αυτά μπορεί να διευκρινιστούν σε επίπεδο 1 όμως οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κάποια ευελιξία όσον αφορά την έκδοση συστάσεων και προσανατολισμών και ερωτήσεων και απαντήσεων για να εξασφαλίζουν εποπτική σύγκληση. Θα βοηθούσε ίσως στον κανονισμό περιποτικών αρχών να θεσπιστεί αρχή της αναλογικότητας και θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να εστιαστούν επ' αυτής της αρχής στην αξιολόγηση συνεπειών για τις ομάδες ενδιαφερομένων κύκλων, stakeholder groups, από την εμπειρία μου σαν πρόεδρος του SMC, να επιχείσω αυτό που είπε η κυρία Φελίθ. Οι ομάδες των ενδιαφερομένων φορέων είναι συμβουλευτική ομάδα κυρίως, αλλά όχι εποπτικός φορέας που εποπτεύει τις εποπτικές αρχές. Συμφωνώ ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να δώσουμε στις ομάδες ενδιαφερομένων το δικαίωμα να αξιολογούν τις κατευθυντήριες γραμμές που ελέγχουν κατά πόσο οι ομάδες των διαφερομένων κινήθηκαν εντός των αρμοδιοτήτων τους ή όχι. Αυτός αλλάζει τους ρόλους, αυτή η προσέγγιση αλλάζει τους ρόλους. Δεν με ικανοποιεί συνεπώ αυτή η σύσταση. Ταυτόχρονα διαβλέπω την ανάγκη για περισσότερους ελέγχους όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων στο τρίτο επίπεδο. Κυρίως όσον αφορά συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο θα, είναι, θα πρέπει να είναι στα χέρια του φορέα εφέσεων ή του δικαστηρίου. Είναι νομικό θέμα κατά πόσο η ΕΣΜΑ κινείται εντός των αρνητήτων της ή όχι. Τώρα για εποπτική σύγκληση και πιο άμεσες εποπτικές εξουσίες. Το ερώτημα της κυρίας Περέζ. Δυσχερέστατη απάντηση. Πρέπει να δεχτώ αρχικά ότι οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη εκτελέσει τα καθήκοντά τους με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά την ΕΣΜΑ, να πω ότι είχε αναπτύξει μια εποπτική μεθοδολογία για την εποπτική σύγκληση. Έχει θεσπίσει αρχές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, των stakeholders, σε αυτό το πλαίσιο και τέσσερα με πέντε χρόνια από όταν εστιάστηκε επί εποπτική συγκλήσεως η ΕΣΜΑ μπορώ να πω ότι πολλά τα επιτεύγματα. Κοινή ε, εποπτική ε, νοοτροπία, η σωστή προσέγγιση έχει θεσπιστεί πλέον και από τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Τώρα χρειάζεται να διαχωριστούν συγκεκριμένα θέματα, ούτως ώστε οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές να μπορούν να εντοπίζουν τα θέματα τα οποία θέλουν να θέσουν στους στόχους. Και μετά βλέπουμε πώς οι εθνικοί φορείς έχουν πετύχει τους εν λόγω στόχους. Συστήνω αυτού, αυτό συγγνώμη, αντί άμεσων εποπτικών εξουσιών, ίσως σε 15-20 χρόνια ε, η ΕΣΜΑ να έχει πιο άμεσες εποπτικές εξουσίες. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε σταδιακά. Προχωράμε και βλέπουμε πώς θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαμπέλα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη. Αν υπάρχει δυνατότητα να αποφευθούν επικαλύψεις μεταξύ εθνικών ελεκτικών αρχών και ΕΣΜΑ. Εγώ δεν διαβλέπω μεγάλο πρόβλημα επικάλυψης και έλλειψης αποτελεσματικότητας. Αν βέβαια η αρχή που διέπει τις λειτουργίες του τομέα είναι μια έσμα που εστιάζεται επί συντονισμού και προθήσεως της εποπτικής συγκλήσεως. Επιπλέον, προφανέστατα βέβαια, υποστηρίζουμε και κάποιες συμπληρωματικές εξουσίες που πρέπει να αντιθούν στην ΕΣΜΑ σε κάποιους τομείς, σε τομείς που δικαιολογείται. Αν περιορίσουμε τις συμπληρωματικές εξουσίες σε κάποιους τομείς και δεν επεκταθούν στα φυλάδια, στους διάφορους, στα διάφορα ταμεία κλπ, θα αποφύγουμε την, ε, το διαχωρισμό και τις ανεπάρκειες ελλείψεις όσον αφορά εποπτική, εποπτεία των ταμείων ή των χειριστικών εταιριών ή ελέγχου των ε, πληροφοριών που διαθέτουν εταιρείε, των περιεχομένων των φυλαδίων κλπ. Αν περιοριστούμε σε αυτά που προτείνουμε, αντί να αυξηθούν οι αρμοδιότητες που ανατίθεται σε αυτούς τους φορείς αν δώσουμε και άλλες ε, αρμοδιότητες για έλεγχο συναλλαγών με χώρες δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι σαν πρόεδρος της Ισπανικής Επιτροπής Αξιογράφων είχα αυτή τη θέση για ένα χρόνο και έχω θετική εντύπωση για την ΕΣΜΑ για αυτά που έκανε μέχρι τώρα η ΕΣΜΑ σε σχέση με την εποπτική σύγκληση, σε σχέση με τη δημιουργία μιας κοινή νοοτροπία και κουλτούρας. Η ΕΣΜΑ είναι ένα φορέα που λειτουργεί καλά. Το πρόβλημα δεν είναι να διορθώσουμε τα κενά και τις αποτυχίες, αλλά να συντονιστούμε με τη φιλοδοξία μας, δηλαδή να πετύχουμε ε, μια ενιαία κεφαλαγορά ευρωπαϊκή και πλήρω πραγματικά ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση όσον αφορά το εποπτικό σύστημα στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί καμιά φορά ε, το, κλίμα είναι κάπως απεσιόδοξο όσον αφορά την ΕΣΜΑ. Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι πολύ καλός φορέας. Και πρέπει να μεγαλώσει και να ισχυροποιηθεί. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τις εκτελεστικές συνεδριάσεις που προτάθησαν για τη μεταρρύθμιση και πώς αυτή η προσέγγιση ταιριάζει με το σύστημα διακυβέρνησης που προτείνεται στα πλαίσια της μεταρρυθμίσεως των ελεκτικών φορέων. Εδώ υπήρξε κάποιο πρόβλημα χρονισμού. Η μεταρρύθμιση του ΕΜΙΡ σχεδιάστηκε παλιά και οι συντάκτες τότε ε, έθεσαν το θέμα αυτών των συνεδριάσεων κλπ. Δεν έχει νόημα αυτό στα πλαίσια της γενικής μεταρρυθμίσεως των ε, φορέων ελέγχου. Εγώ θα έθετα τις ευθύνες για τους ελεγκτικούς φορείς εντός του Διοικητικού Συμβουλίου. Και η ιδέα, σύμφωνα την οποία ένα από τα μέλη έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την εποπτεία των CCPs που αποστολεί αυτού είναι πάντα να εξετάσει αυτή την πτυχή, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Όσον αφορά τα φυλάδια, ποιο ήταν το ερώτημα, πώς να πετύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση στον τομέα. Τα εφιστάμενα εργαλεία, εάν ενισχυθούν και βελτιωθούν μάλιστα, ίσως να αρκούν και με το παραπάνω εξέταση ομοτήμων, Φερρυπίν, τον οποίο θα ηγείται η ΕΣΜΑ. Το εργαλείο της παραβιάσεως του δικαίου που χρησιμοποιήθηκε σπανίως μέχρι τώρα και κάτι άλλο έχω υπόψη μου το άλλο εργαλείο για εποπτικό σχεδιασμό και αυτό μπορεί να είναι χρησιμότατο. Και βέβαια, εκρεμεί ακόμα το θέμα της εφαρμογής των μέτρων επίπεδου 2 και 3, δυνάμει του νέου κανονισμού περί φυλαδίων. Και ίσως αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι όλα ρυθμίζονται παρκώς και να αποφύγουμε ε, ρυθμιστική διατησία σε αυτά τα επίπεδα. Αυτά και ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο από τη Finance Watch. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Έχουμε την ομάδα των εμπλεκόμενων φορέων και ύστερα το θέμα τη εντολή τη προστασία των καταναλωτών σε ό,τι αφορά του εμπλεκόμενου φορεί, τα ενδιαφεραμένα μέρη, σε ό,τι αφορά και αυτά που είπε ο κύριος Βέλτσε. Πρόκειται για ομάδες οι οποίες έχουν ε, συμβουλευτικό καθαρά ρόλο και το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ προσωπικά είμαι μέλος της ομάδας ε, των τραπεζικών αρχών της Ευρώπης. Ε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος τη δράση των ομάδων αυτών. Να απαντούμε σε ερωτήσεις, κάνουμε προτάσει πρωτοβουλία, προτείνουμε διάφορα θέματα και πρόκειται για ένα είδος, αν θέλετε, καταπιστεύματος, αλλά σε πολύ απλούς όρους δεν βλέπουμε να έχει αλλάχθει οποιαδήποτε αλλαγή κειμένου, να μην υπάρχει, δεν έχει υπάρξει δηλαδή οποιαδήποτε αντίκτυπο τη δουλειά της ομάδας των ε, stakeholders. Αυτό που θα μπορούσε λοιπόν να αλλάξει θα ήταν η υποχρέωση όπως υπάρχει σε κάποια πάνελ καταναλωτών που έχουν συσταθεί σε κάποιες χώρες προκειμένου κάθε, κάθε αρχή να υποχρεούται να απαντήσει στα σχόλια που έχουν γίνει από την ομάδα αυτή των εμπλεκόμενων φορέων. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση, τη σύνθεση τώρα, είναι σημαντικό να είναι πραγματικά ισόρροπη. Σαφώς υπάρχει ανισορροπία μεταξύ τους εκπροσώπους ε, της βιομηχανίας και των χρηστών. Ε, σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους της βιομηχανίας του κλάδου βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία προετοιμάζουν τις παρεμβάσει του που κάνουν μια δουλειά η οποία δεν ε, προβάλλεται στις συναντήσεις. Ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά την ομάδα των χρηστών. Άρα, δεν πρόκειται για αποζημίωση για τους χρήστες, για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, για τα συνδικάτα. Πώς αποζημιώνουμε τις ομάδες αυτές για τον χρόνο που δαπανούν. Θα μπορούσαμε να θα ορίσουμε και μία χρηματοδότηση για τους εκπροσώπους των χρηστών για να μπορούν να κάνουν επιπλέον έρευνα. Για το θέμα της εντολής προστασίας ε, των χρηστών των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως θα γνωρίζετε, η Finance Watch μαζί με άλλους ε, εκπροσώπους των καταναλωτών, των ε, οικογενειακών επιχειρήσεων, μικρών επενδυτών έχουν εκφράσει η μεγάλη τους απογοήτευση σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση, την πρόταση αναθεώρησης ε, του κανονισμού, γιατί το σκέλος προστασίας του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις τρεις εποπτικές αρχές είναι πολύ περιορισμένο στην, δημο... Ε, στην Πέρσι, στην διαβούλευση που έγινε μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρήσαμε ότι υπήρχε μια πρόθεση να αυξηθεί ε, αυτή η προστασία σε ό,τι αφορά και το μοντέλο Twin Peak, σε ό,τι αφορά δηλαδή την επιχειρηματική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε σε καμία περίπτωση στην πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού. Θα θυμάστε θα ήταν να ανατεθούν ε, αυτές οι αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Θα ήταν τεράστιο μα, βήμα αυτό για μας. Φυσικά θα προτιμούσαμε να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή αρχή, αλλά τουλάχιστον θα ήταν ένα μεγάλο βήμα, μεγάλη πρόοδος να ανατίθενταν αυτές οι αρμοδιότητες στην ΕΣΜΑ. Αν παραμείνει αυτό σε επίπεδο εθνικών αρχών προστασίας του καταναλωτή, αυτό θα αποτελούσε, να το θέσω αλλιώ, το κατώτατο όριο, το ελάχιστο όριο για μα, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα θετία. Κατ' ελάχιστον, λοιπόν, θα θέλαμε να μπει στο κείμενο ότι θα δοθεί χρηματοδότηση προς τον ε, σκοπό αυτό. Ιδάλλως θα παραμείνει ακόμα υπό του ραντάρ. Σε ό,τι αφορά τις υποπτικές αρχές, δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Σούφελτ λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάφορα ζητήματα παρουσιάστηκαν και να ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Μπάλτς για την αναλογικότητα. Η αναλογικότητα όντως αποτελεί μία από τις ε, πιο βασικές αρχές σε διαφορά τις δραστηριότητες αυτές κατά τη γνώμη μου, στηρίζεται σε διάφορους πυλώνες η αναλογικότητα. Καταρχάς, η νομική διαδικασία, όπως την περιέγραψε και ο κ. Βέιλ. Αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, όσο πιο πολύ η πολιτική παραμένουν με ευρείες νομικές έννοιες, το οποίο αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, τόσο πιο πολύ υπάρχει ανάγκη διευκρίνηση. Ιδάλω, πώ θα γίνει η υλοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει δεύτερο και τρίτο επίπεδο, λοιπόν. Η αναλογικότητα, λοιπόν, θα ήταν διαφορετική εντελώ αν ε, υπήρχε πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση σε πρώτο επίπεδο. Αλλά ακόμα και αν δεν γινόταν αυτόν, σε καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ρύθμιση σε πρώτο επίπεδο. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό και αποδεκτό και απαραίτητο να υπάρχει διευκρίνηση. Διευκρίνηση των... σε διοικητικό επίπεδο. Επαναλαμβάνω και θα ήθελα να προασπιστώ την συμπεριφορά των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών σε ό,τι αφορά το τρίτο επίπεδο. Γιατί χρησιμοποιήθηκε ο όρος self-empowerment. Οποιαδήποτε αρχή που έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν, που δεν υποχρεούται να εξηγήσει το πώς εκτελεί αυτά τα καθήκοντα δεν έχει αυτό το self-empowerment. Φυσικά μπορεί να υπάρχει το ερώτημα και το θέμα της υπέρβασης των αρμοδιοτήτων αυτού και συμφωνώ με τον κύριο Βάιλ, πρέπει να ελέγχεται και ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές στις οποίες μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φορέα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το, Γενικό Δικαστήριο θα μπορούσαν να είναι αρμόδια και ενδεχομένως να βοηθούσε και ένα Δυτικό δικαστήριο. Ένα άλλο στοιχείο της αναλογικότητας είναι η διάκριση της ρυθμίσης και της εποπτείας. Η εποπτεία θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο επίπεδο κατάρτιση τη νομοθεσία, γιατί πολύ απλά δεν θα κάνει αλλιώ τη δουλειά τη. Όσο πιο πολύ απέχουμε και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση ενό ιστορικού πειράματο σε ό,τι αφορά την τραπεζική εποπτεία στην Ευρώπη. Σε επίπεδο έχει πλέον ε, φτάσει αυτή η εποπτεία. Προσπάθησα την προηγούμενη εβδομάδα να κοιτάξουμε πώς μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο λεπτομέρειας για τις μεμονωμένες ευρωπαϊκές τράπεζες. Είναι τεράστια η πρόκληση. Θα πρέπει η εποπτεία να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρωτογενές επίπεδο για να υπάρχει αναλογικότητα. Να αναφερθώ τώρα σε κάποιες βασικές, ε, σε κάποια, σε κάποια σημεία ορολογίας. Ε, σύγκληση, υποπτική σύγκληση, διακυβέρνηση, είπε η και να αποφευθεί ο εποπτεύον του εποπτεύοντος. Η εποπτική σύγκληση προφανώς είναι σημείο κλειδί σε ό,τι αφορά τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία των εργασιών τους. Θα ήθελα, μάλλον σε αντίθεση με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, μου κάνει κάπως εντύπωση ο βαθμός σκεπτικισμού από πλευράς κάποιων ευρωπαϊκών εκπροσώπων σε ό,τι αφορά την επιτυχία που είχαν σημειώσει ως τώρα οι Ευρωπαϊκές Επιτροπικές Αρχές. Εγώ έχω να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ευρωπαϊκές Αρχές, οι Επιτροπικές Αρχές κάνουν εξαιρετικό έργο, πάρα πολύ σημαντικό και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να πιέσουμε μία λύση, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν βασμία, σταδιακά. Ένας κώδικα σχετικό έχει δημιουργηθεί και στις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και θα πρέπει να ακολουθηθεί και στο μέλλον αυτή η προσέγγιση μου. Θέσατε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Τι πιστεύω για τις εθνικές εποπτικές αρχές σε περίπτωση που δεν κάνουν τη δουλειά τους και κατά πόσον οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα μπορούν να παρέμβουν. Ναι, θα πρέπει, αλλά το κάνουν και όλα ήδη. Σήμερα έχουν σχετική εντολή. Και εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοιε συζητήσει σε διάφορες περιστάσεις. Εγώ ο ίδιο δεν έχει ακόμα χρειαστεί, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δυνατότητα αν πραγματικά χρειαζόταν. Πριν από κάποιες εβδομάδες με το MIFID και το MI4 ε, εισήχθη ένα τελείως καινούριο πεδίο αρμοδιοτήτων. Υποθέτω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά στην πράξη. Άρα δεν... Ε, αυτό που δικαίως ρωτάτε για τις επικουρικές αρμοδιότητες από πλευράς των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Πιστεύω ότι είναι δεδομένο σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση, το governance. Ε, για να κλείσω στο σημείο αυτό να αναφέρω Κάτι που είπε και ο κ. Λιντελαρουζιέρ και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και να μην το παραβλέπουμε. Ενδεχομένω είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίζονται όλε οι ευρωπαϊκέ υπηρετικέ αρχέ με τον ίδιο τρόπο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ενδεχομένω ότι προχωρούν προ τα εμπρό, προοδεύουν, αλλά στην πορεία αυτή θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση. Τι να δημιουργηθούν ε, ευρωπαϊκές υποπτικές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών δεν έχει νόημα στην ΑΙΟΠΑ. Έχετε ε, δίκιο, κύριε Ντελαροζιέρ, ε, για τα ιστορικά μοντέλα, αυτό που είπατε. Δεν έχει νόημα πάλι να δημιουργηθούν ιστορικέ δομέ. Η ΕΣΜΑ, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, είναι διαφορετική περίπτωση. Ο κ. Αλμπέλα είπε ότι λόγω πρακτικών ρυθμίσεων δεν έχει... Δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις πολύ λεπτομερείς. Ε. Άρα εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα και πάλι θα αναφέρω αυτό που είπε ο κύριος Λαροζιέρ. Συμφωνώ απόλυτα. Θα προτιμούσα ένα μοντέλο όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποκαλυφθεί εκτελεστική επιτροπή και να έχουμε δύο, τρία, τέσσερα πλήρη μέλη που θα έχουν εποπτικές αρμοδιότητες. Αυτό θα είχε νόημα αν δεν εμποτίζεται στο έργο της η Επιτροπή Εποπτών. Αν ε, σωστά κατάλαβα και εσείς συνάδελφε το θέσατε το θέμα αυτό. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΣΜΑ θα δημιουργούσαμε μια τριπλή ε, δομή μια τριπλή δομή και αυτό με όλο το σεβασμό που σας τρέφω δεν έχει νόημα και θα ήθελα να το αποφύγουμε. Άρα, εγώ θα προτιμούσα αυτό που είπε ο κύριος Λαροζιέρε, γιατί αποτελεί μια πρακτική προσέγγιση η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη διαφοροποίησης μεγαλύτερης μεταξύ της εποπτείας και της διακυβέρνησης. Τελευταία ερώτηση για την χρηματοδότηση, κυρία Μπερές. Ναι, όντως, σύμφωνα με τη λογική που πρότεινα, είναι αποδεκτό και αποτελεί αυτό μάλιστα κοινή πρακτική, να σας πω, παντού. Να υπάρχουν εισφορές των εποπτευομένων οργάνων για την εποπτεία. Και άκουσα με προσοχή τον κύριο Λαροζιαρ γιατί αυτό που είπε για τη πρόταση του 60% είχε να κάνει με το βαθμό στον οποίο ασκούν υποπτικές αρμοδιότητες ε, οι υποπτικές αρχές. Αυτό ισχύει για την ΕΣΜΑ, αλλά όχι για τις άλλες δύο αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Και όντω, κάποιοι από εμά ε, ε, πλαγήκαμε όταν ακούσαμε ότι θα ήταν μια μόνη μεγάλη πρόταση. Ε, αυτά. Ο Ζακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν. Καταρχάς από τον κύριο Μπάλτσα. Πιστεύω ότι όταν κανείς θέλει να κατανοήσει την ουσία του τι χρειαζόμαστε ως προς τη διακυβέρνηση, αυτή ήταν η ερώτησή σας, πρέπει να σκεφτεί κάτι πολύ απλό. Ε, βασικά, αρχικά σκεφτήκαμε τη ρύθμιση, γιατί πραγματικά μας έκανε ε, να φρικιάσουμε το ότι υπήρχαν τόσοι διαφορετικοί κανονισμοί από τη μία χώρα στην άλλη. Οπότε ε, δώσαμε την έμφαση σε, μία μόνη, σε ένα μόνο εγχειρίδιο, σε έναν μόνο κανονισμό για να, που θα ισχύει για όλους και θα τελειώνουμε. Αλλά πιστεύω πως οι τρεις ΕΖΑ καλά έκαναν και το σκέφτηκαν αυτό αρχικά. Όμως καθώς περνά ο καιρός και βλέπεις ότι όντως έχεις έναν ε, τέτοιο νέο βιβλίο, ε, διαπιστώνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις όλα αυτά στην πράξη. Και γι' αυτό και υπερβάνω και δικαίως ε, τόνισε την σύγκληση της εποπτείας. Οπότε, πέρασε αυτή η ε, ιδέα από τους περισσότερους κοινού κανόνες σε μεγαλύτερη σύγκληση των υπερχόντων κανόνων. Γιατί υπάρχουν άλλες χώρες που το εφαρμόζουν ε, έτσι, άλλες αλλιώς, οπότε είναι περίπλοκο το θέμα και πιστεύω, όπως ε, θύμισε μόλις και ο κύριος Χούφελ, ότι Μπορούμε καλύτερα να το προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα της σύγκλησης στην εποπτεία εάν εάν αν ενισχύσουμε το, το Διοικητικό Συμβούλιο με ανθρώπους που είναι αδιαφεσβήτητοι, που έχουν δείξει δηλαδή με την πορεία τους ότι γνωρίζουν αυτό αυτά τα προβλήματα, ότι είναι αντικειμενικοί. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ε, και ε, νομίζω πως ε, θα ήταν θετικό κάτι τέτοιο. Γιατί αν μπει κανεί σε μια σύγκρουση συμφερόντων και έχουμε και εκπροσώπηση αυτών στο Εποπτικό Συμβούλιο, πολύ δύσκολο. Γιατί όπως δεν θέλουμε να πληγώσουμε κανέναν, θα πιστεύουμε ότι ε, θα είναι ικανοποιητική η κατάσταση διαφορετικά, οι επικρίσει είναι πολύ πιο εύκολε. σε πάση περιπτώσει μπαίνει σε ένα δύσκολο πλαίσιο. Ενώ αν έχεις δύο-τρει ανθρώπους οι οποίοι είναι ανδιαφυσβήτητα κορυφές σε αυτό το, στον τομέα τους, νομίζω πω αυτό θα ήταν πολύ θετικό, όχι μόνο για την λόγο εποπτική αρχή, αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα, γιατί εν τέλει εσείς στο Κοινοβούλιο έχετε αποφασίσει για αυτά τα θέματα σύγκλησης. Οπότε πρέπει να εφαρμοστούν και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την θετική και αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος θα ήταν θετικό. Για την Φλωράνς Μπερέζ, ε, περβάζω διορθώνει ο μιλητής Μπερέζ, ε, ρωτήσατε δύο θέματα. Ε, καταρχάς, ε, η ιδέα της ύπαρξης ενός ειδικού για τα CCPs στα Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό που λέω. Ε, καλή ιδέα. Δεν είναι ποτέ κακή ιδέα να έχεις κάποιον που ξέρει τι λέει. και θα συμφωνούσα. Θα διαφωνήσω με μία πτυχή των προτάσεων της Κομισιόν που λέει ότι θα πρέπει να δικαιωθεί ένα υποσυμβούλιο για τα CCPs. Νομίζω πως αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό. Και προτιμώ τη δική σας πρόταση. Και έπειτα, ε, με ρωτήσατε κάτι για την, ε, για την ESRB. Πρέπει να παραδεχτώ ότι κάναμε ένα ασφάλμα όταν ε, συντάξαμε αυτή την έκθεση. Δεδομένου στις καθεστέρες τη ΕΚΤ που έχει μεγαλύτερο κύρος, περισσότερη ε, αξιοπιστία κτλ. Το έργο της μικροεποπτείας Και διαπίστωσα μετά ότι δεν ήταν τόσο καλή ιδέα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ρωτήσουμε από την ΕΚΤ να ζητήσουμε μάλλον από την ΕΚΤ αν μία, ένας μάλλον ε, κατά κάποιο τρόπο οργανισμός, αν μπορεί να φτιάξει και να ασκήσει δική τη ε, ε, πολιτική νομισματική και αυτό θα μπορούσε να διαταράξει τις αγορές Ο δυναμισμός ε, ε, ενό τέτοιου οργανισμού είναι πολύ χαμηλός και η αποτελεσματικότητά του στις αγορές ε, είναι σχεδόν μηδενική. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλύτερη ιδέα εδώ να έχουμε μια SRB που θα είναι λίγο πιο απομακρυσμένη από την ΕΚΤ που επίσης θα έχει ε, πανεπιστημιακού επίπεδου προσωπικό μεγάλου κύρους ε, που είναι δεν θα έχει αρμοδιότητες, αλλά θα είναι η αρχή η οποία θα βαραίνει στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν ε, οι κυβερνήσεις αυτήν την υπόθεση. Και κάτι που είπε η Περβάνος και που είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για την για την Ένωση των Κεφαλαίων Κατά τη γνώμη μου η ΕΣΜΑ που δεν θα πρέπει να διαταράσσεται από πολλές ε, ε, αρμοδιότητες, περιτές κτλ. Ε, Η ιδέα λοιπόν είναι ότι έχει σπουδαίο μέλλον. Γιατί, γιατί μετά από θα καταλαγιάσει η, ε, ε, το Brexit, ε, τα, οι συνέπειες μάλλον του Brexit, θα έχουμε την Ελβετία και Ποιος θα είναι σε θέση να φτιάξει μία πλατφόρμα συνεργασίας στην Ευρώπη που θα εξετάσει το μέλλον εκείνης της ευρωπαϊκής αγοράς στον πραγματικό κόσμο που είναι παγκοσμιοποιημένος και απάντηση είναι είτε θα το κάνει η παλαιά διπλωματία του 19ου αιώνα όπου η τράπεζα της Αγγλίας ε, τσακώνεται με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε θα είναι μια διαδικασία συνεργασίας. Και αν είναι διαδικασία συνεργασίας, όπως εγώ τουλάχιστον θα ήθελα, η ΕΣΜΑ θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο εκεί. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ΕΣΜΑ. Δεν θα πρέπει να την πιέζουμε υπερβολικά σε πολλά νέα πράγματα. Βήμα το βήμα, όπως άκουσα από τον φίλο εξ αριστερών, είναι αυτό που θέλω κι εγώ και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που δημιουργήσαμε το 2010-2011 με τη ΣΕΣΜΑ θα αποκτήσει όλα ένα και μεγαλύτερη σημασία και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. με του Σκιώδης και το Κατζιάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, η κυρία Σουενμπόρνα. Σας ευχαριστούμε για τα σοφά σας λόγια που σίγουρα θα τα πάρουμε όλοι ε, σοβαρά υπόψη. Να σας τονίσω, επίση να σας ευχαριστήσω μάλλον ε, που ε, περάσαμε αυτή την, ΕΣΑ, ε, την νομοθεσία περί ΕΣΑ, περί υποπτικής αρχής εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο είμαστε πολύ περήφανοι. Έχουμε επικριθεί βέβαια, αλλά όντως λειτουργούν και έχουν και ε, Κοινού κανόνε Βέβαια έχουν αποκλείσει. Εγώ εργάζομαι με την ΕΣΜΑ και την ε, αγορά στην εργασία τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ περισσότερο. Ε, αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ένα από τους προτείνει ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να δίνουν περισσότερε λεπτομέρειε στα επίπεδα 1, 2, 3. Ενώ εμείς προσπαθούμε αυτό να το αναθέσουμε στου ειδικού και όχι στους πολιτικούς. Ε, πού είναι η ισορροπία λοιπόν σε όλα αυτά. Εμείς είμαστε αρκετά εμπειρογνώμονες για να κάνουμε πιο λεπτομερή δουλειά από ό,τι κάνουμε. Και έπειτα για τη σύγκληση. Δεύτερος μεγάλος ρόλος που ανέλαβαν η ΕΣΜΑ και άλλες εποπτικές αρχές είναι αυτό τη σύγκληση. Το μοντέλο για τη σύγκληση έχουν φτιαχτεί. έχει φτιαχτεί και τα εργαλεία. Το θέμα είναι όμως ε, χρησιμοποιούνται. Έχουμε τα μητρώα ε, ε, ας πούμε σε έξι ε, τέτοια μητρώλα εκεί λειτουργούν τα τέσσερα και όχι τα δύο. παρότι είχαν αρκετό χρόνο για να τα θέσουν όλα αυτά σε εφαρμογή. Το θέμα της τυποποίησης είναι επίσης πολύ σημαντικό. Για τη ΜΥΦΙΤ 2 επίσης, πώς στάσαμε σε αυτό το στάδιο ώστε η βασική μας νομοθεσία για τις αγορές καθυστέρησε ένα χρόνο και 17 κράτη-μέλη δεν την είχαν μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία. Ένα χρόνο μετά. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό, δεδομένου το τι συζητάμε με τις εθνικές αρχές ε, καθημερινά. Η ιδέα ότι ξέφυγαν ε, ε, χωρίς καμία τιμωρία και ενώ δεν το εφάρμοσαν ε, και λένε ήδη ότι α, δεν πρόκειται να λειτουργήσει, θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Και έπειτα, η άμεση εποπτεία των CCP είναι πολύ πολιτικοποιημένο θέμα και πολύ επίκαιρο. Εγώ τα τελευταία νέα χρόνια εργάζομαι για τα, με, εμπορικά, με τα ε, επιρροές στις αγορές και τα CCP και τα CDT εφόσον, η, εφόσον λοιπόν συμφωνούμε ότι τα CCP πρέπει να εποπτεύονται από την ε, εποπτική αρχή. Γιατί όχι και τα CSD, εφόσον ξέρουμε ότι το ICSD είναι αυτό το οποίο ε, παρέχει την άμεση δυνατότητα μεταφοράς των πολιτικών στην αγορά. Να μην βλέπουμε λοιπόν μόνο τα επίκαιρα ε, CCP, ε, επειδή αυτά έχουν πάρει πολιτικό χαρακτήρα αυτού του είδους η συζήτηση μετά το Brexit. Έπειτα, συστημικά σημαντικά CCP υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να... Ε, και έχουμε εδώ τον επόπτη ε, κάνουν εξαιρετική δουλειά, φανταστική δουλειά με την συγκεκριμένη ε, μονάδα. Γιατί η ΕΣΜΑ θα κάνει κάτι καλύτερο. Ανησυχώ λοιπόν κάπως για το ρόλο της ΕΣΜΑ, εφόσον έχουμε πολύ ικανούς υπόπτες που κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα. Και ένα σχόλιο για σχέση, σε σχέση με το φυλάδια ε, Υπάρχει όλα είναι και μεγαλύτερη ανησυχία πως ίσως αυτό δεν χρειάζεται να γίνει και να περάσει από έγκριση στην ΕΣΜΑ. Και σίγουρα όταν εγώ έκανα την νομοθεσία τη σχετική πρόσφατα, πρόκειται για ένα, μια νομοθεσία, ένα κανονισμό, το συζητήσαμε πάρα πολύ καιρό και αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να είναι εντολή τη ΕΣΜΑ. Το θέμα είναι όμω ότι σε κάποια από τα γεύματα εδώ στα κοινοβούλια το χρηματιστήριο του Λονδίνου, μάλλον ο γενικό διευθυντή του Χρηματιστήριου του Λονδίνου, είπε ότι από όλου του δείκτε του LSE ούτε μία μονάδα δεν χρησιμοποιεί το διαβατήριο για το προσπέκτους. Άρα λοιπόν τι προσπαθούμε να δείξουμε, να δώσουμε μάλλον στην ΕΣΜΑ να αναλάβει εφόσον δεν υπάρχει δραστηριότητα γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι αγωγής έχω να πω κάτι και μετά έχω ρωτήσεις. Όλοι συμφωνούμε περιστόχων, Καλύτερη υποπτική σύγκληση, εξάλληψη τρευλώσεων και ρυθμιστικής διατησίας και επίπεδο προστασίας για τον κατανοτή ψηλό και παρόμοιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν αποτελεσματικά. Αναφέρθηκε ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί εξελικτικά 10 με 15 χρόνια αναφέρθηκε σαν περιοδο εχουμε Έχουμε 10-15 χρόνια. Δεν ξέρω. Ο τομέας χρηματοστατικών ε, συναλλαγών αναπτύσσεται τάχιστα στην Ιφίλιο, κυρίω στην ε, Ασία. Και λόγω νέα τεχνολογία ίσω να υπάρχουν φορεί και παίκτε στην αγορά που θα παρουσιαστούν που δεν του ξέρουμε σήμερα. Και θα καταφτάσουν τάχιστα και αυτοί δεν θα υπόκεινται στο παραδοσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην ύπαρξη χρόνου. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Στις ερωτήσεις τώρα. Για το πρόεδρο του Μπάφιν που είπε ότι δεν θέλουμε επόπτη το επόπτη. Συμφωνώ με αυτό. Ερώτηση. Διαβλέπετε κάποιο κίνδυνο αν εφαρμόσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπευλήθη ότι αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε εχθρική αντίδραση κυρίως από πλευράς εκείνων των φορέων των ελεκτικών που είναι καλά εξοπλισμένοι όπως είναι EMF, Buffin κλπ. Μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο σαμποτάζ, δολιοφθοράς της επικοδομητικής συνεργασίας, κάτι άλλο. Απ' την άλλη, πρόσφατα, στη Λετωνία είχαμε υπόθεση. Η τράπεζα EBLB χρεοκόπησε και έγινε καθάριση. Ερώτηση. Πώς γίνεται η Εθνική Αρμόδια Αρχή της Λετωνίας και οι ελεγκτικοί φορείς οι άλλοι ευρωπαϊκοί να μην βλέπουν αυτή την εξέλιξη. Τι θα έπρεπε να αλλάξει για να μην εμφανιστεί ένα παρόμοιο φαινόμενο και μάλιστα σύντομα. Δεύτερη ερώτηση. Στον εκπρόσωπο της Finwatch. Αφορά τη χρηματοδότηση η ερώτηση. Προτάθηκε από τον πρόεδρο του Μπάφη να κάνουμε διάκριση μεταξύ ρυθμιστικών ταμείων και ποπτικής χρηματοδοτήσεως. Ερώτηση. Η Finwatch τι λέει αυτό. Η Financial Watch. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Έχει νόημα να εξαλειφθεί η οικονομική συνεισφορά των εθνικών ελεγκτικών φορέων. Εγώ το αμφισβητώ προσωπικά. Θα ήθελα να παραμείνουν οι εθνικοί φορείς ελέγχου στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεως της ΕΣΑ. Αν διαχωριστεί χρηματοδότηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως 40% και των υπολείπων που θα προέρχονται από τον χρηματοδοτικό τομέα, τι διαβλέπω, ότι δεν θα ελέγχονται οι δραστηριότητες αποτελεσματικά και θα έχουμε υψηλό κόστος αδικαιολόγητο. Τρίτη ερώτηση. Κύριε Ντελαγοζιέρ, για το ESRB. Κατά πόσο τα ESRBs θα πρέπει να έχουν την ίδια προεδρία. Το συζήτησα πρόσφατα. Και τι διαπίστωσα άκουσα να μου λένε ότι είναι ένα μαύρο κουτί τα ECRB. Και δεν επικοινωνεί το ECRB με τον έξω κόσμο όσον αφορά το τι κάνει και πώς το κάνει. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους και μεθόδους δυσνοήτους ε, για όλους τους άλλους. Όλοι αγνοούν τις λεπτομέρειες. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Τι προτείνεται. Ούτως ώστε η συνεισφορά του ECRB ε, να είναι θετική και να γίνει αντιληπτή ως τέτοια. Αυτά και ευχαριστώ. Σπεν Γκίγκολτ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγιναν στα πλαίσια εκθέσεως του Κοινοβουλίου της πρώτερης θητείας. Εγώ είχα γηθεί των εργασιών τότε. Και σε ένα πόρισμα συμφωνήσαμε. Κάτι που ακροθυγώς αναφέρθηκε. Ποιο είναι το βασικό αυτό πόρισμα. Όταν δημιουργήσαμε τους Εθνικούς Φορείς Ελέγχου, δώσαμε σαφή εντολή. Αρκετά ευρία εντολή. Και γι' αυτό η συζήτηση κατά πόσο ξεπεράστηκε η εντολή θεωρώ ότι είναι αστεία. Θα ήθελα ένα παράδειγμα να μου δώσετε. Πού παρέβησαν την εντολή τους ε, οι εθνικοί φορεί. σύμφωνα με τον κύριο Ούφελτ. Όταν το έθεσε αυτό, κανείς δεν μου έδωσε παράδειγμα. Και τελώνει αναμονή ακόμα. Πέραν αυτό. Δώσαμε αυτή την ευρεία εντολή. Βλέποντας τι έκαναν οι φορείς ελέγχου, τι εξουσίες χρησιμοποίησαν, βλέπουμε ότι υπάρχουν τομείς όπου έκαναν πολλά μπήκαν σε λεπτομέρειες, δεν κινήθηκαν επαρκώς αναλογικά και συμφωνώ σε κάποιο βαθμό με αυτό. Όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων, οι εθνικοί φορείς τα πήγανε μια χαρά. Όμως, αν ρωτήσεις τους καταναλωτές και τις εταιρείε χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών και τους πεις αισθάνεστε ότι είναι δίκαιοι οι κανόνες και οι όροι που επικρατούσαμε στην Ευρώπη. Υπάρχει ισότητα όσον αφορά την εποπτεία και όσον αφορά τη λειτουργία των διαφόρων αγορών για πλευρά ζήτηση και προσφοράς. Θα μας πούν όχι, πόρα απέχουμε από τους στόχους ε, της ε, ενώσεως κεφαλαγορών. Και αυτό διότι οι εθνικοί φορείς ελέγχου δεν χρησιμοποίησαν όλες τις διαθέσιμες εξουσίες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες τις εξουσίες, αλλά σημαντικότερη είναι η παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και η πρόθεση κοινή νοοτροπία εποπτεία. Άρα, ερώτηση προ το πάνελ. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνετε ούτω ώστε να τεθεί τέρμα στη μη εφαρμογή και μη χρήση των αντιστοίχων εξουσιών και στόχων. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Δηλαδή ακόμα οι απλοί καταναλωτές πληρώνουν πολύ ψηλά ποσά για πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουν. Τελευταία ερώτηση του κ. Ντελαροζιέρ. Κατά την άποψή μου, κάνατε μια πολύ καλή πρόταση όσον αφορά τη διοικητική δομή των εθνικών φορέων εποπτεία. Και με την αυτοκριτική σας που εκφράσατε και συμφωνώ μαζί σας ως Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατασκευή, την οικοδόμηση του ECRB. Αλλά αν βγει το ECRB εκτός ΕΚΤ ή αποκτήσει άλλο πρόεδρο, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του ανέφερε Βόλφ Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κοινός καθορισμός ευθυνών. Έχουμε τεράστιο, τεράστιες εξουσίες του Προέδρου και ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων την, α, αποφάσεις. Αν είχαμε πιο μικρό διοικητικό φορέα στην ECRB, αποτελούμενο από επιφανείς ειδικού μακροοικονομικής σταθερότητας και θα είναι ένα συμβούλιο ουσιαστικά οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη, όπου εκεί μπορούν να επιμεριστούν οι ευθύνε. Σαφώ να οριοθετηθούν οι ευθύνε. Και μετά, αυτό ο φορέα συνεργάζεται με ευρύτερη ομάδα μελών, όπω ισχύει τώρα, στο παρόν η CRB. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λάγκεν έχει το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να κάνω δύο μικρές ερωτήσεις ε, το ένα είναι η κρίση στη Λετωνία. Εδώ θέλω να ακούσω την άποψη των ειδικών. Κατά πόσον ε, η, υπηρεσία, η αρχή τραπεζών και η ΕΣΜΑ μπορεί να επιβεβαιώσουν την κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση για το μέλλον. Το δεύτερο είναι το θέμα της δυνατότητας του να θέτουμε εμείς, ε, να θέτουν οι ίδιες θέματα είπε ο συνάδελφος Γκίκολντα ότι μόνο ένα παράδειγμα έχει να αναφέρει όπου οι, Ευρωπαϊκέ επαπτικέ Ευρωπαϊκές Αρχές ε, έχουν κάνει μια πρόταση πέρα από την εντολή τους, αλλά η ΙΟΠΑ ξέρω ότι έχει πολλές, σε πολλές περιπτώσεις κάνει κάτι τέτοιο. Για προτάσεις το που δεν ε, είχαν ε, πλειοψηφία για το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποια είναι η άποψη των ε, ειδικών για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Σαΐς. Σας ευχαριστώ πολύ για την συντομία. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, για την συνεισφορά του στη σημερινή συζήτηση και μου έκανε εντύπωση και αυτό που είπε ο κ. Τράκη χθε, μιλώντα για την κρίση, ότι δεν ήταν ε, στην ουσία τη τραπεζική κρίση. Ότι ήταν ε, αποτυχία της ρύθμισης και της υποπτίας. Αυτές λοιπόν οι προαπαιτήσεις, οι εποπτεία και η ρύθμιση θα πρέπει να συντονιστούν για να επιτευχθεί επιτυχία, αλλά με ένα λογικό τρόπο. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ένωση κεφαλαγορών που θα έχει νόημα και κυρίω. Σημειώνω αυτό που είπαμε και για το Brexit. Τι είδου καταγερματισμό θα μπορούσε να αποτελέσει απόρρια του Brexit. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την ε, οικονομική σταθερότητά μας. Να μην το υποτιμούμε λοιπόν αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Όταν ε, ήμουν υπεύθυνο για το φάκελο ΑΙΟΠΑ, είναι σημαντικό γιατί είδα τη σημασία μάλλον της αρχής, γιατί είναι ε, διαμεσολαβητής ε, ουσιαστικά η ΑΙΟΠΑ και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διασυνοριακή αγορά λειτουργεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα όπου δεν λειτουργεί αυτή η διασυνοριακή αγορά, ακριβώς ε, επειδή είναι επιθετική η προσέγγιση των ε, ρυθμιστικών αρχών έναντι των άλλων ρυθμιστικών αρχών και θεωρώ ότι υποτιμούμε σε σχέση με αυτά που είπε ο Σβέν σε ό,τι αφορά την κοινή κουλτούρα εποπτείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έρχονται σε μία τράπεζα και να συναντιόνται οι εποπτικές αρχές για να διευκρινίζουν πολλά από τα ζητήματα για να βρίσκουν τις καλύτερες πρακτικές για να εντοπίσουν περιπτώσει κατάχρηση τη ε, ενιαία αγορά και να μπορούν να θέσουν κοινού στόχου στην εποπτεία. Και για να συμφωνήσω και με τον κύριο Λάγκε, να πω ότι έχουμε δει παραδείγματα υπέρβαση των αρμοδιοτήτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νομοθεσία που έχει προτείνει το Κοινοβούλιο. Και είδαμε πρόθεση ναι. πρόσφατα νομοθεσία σε ό,τι αφορά την κατάργηση με το χώρο εντελώς αντίθετη με αυτά που είχαμε συμφωνήσει και με την συζήτηση που έγινε μετά. Και το είδαμε και στην περίπτωση των προσπέκτους. Ε, όπως είπε η Κέιτ έχουμε δει παραδείγματα όπου υπάρχει υπέρβαση καθηκόντων και σε ό,τι αφορά πρόσφατα θέματα που έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Η συγκεκριμένη λοιπόν ερώτηση που έχω να κάνω σε ό,τι αφορά τους πόρους. Η μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, νομίζω ότι υποτίμησε τις επιπλέον ανάγκε ανάγκες προσωπικού και σε ό,τι αφορά την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του προσωπικού. Και οι απόψεις της αντιπροσωπείας μου είναι γνωστές. Εγώ είμαι ε, κατά τη πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μήπως έχουμε υποτιμήσει σημαντικά τον αριθμό και το επίπεδο των ανθρώπων που χρειαζόμαστε για να εκτελεστούν αυτές οι επιπλέον ε, αρμοδιότητες που αναφέρονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση για τους ε, ομιλητές. Παρατήρηση ταυτόχρονα και ερώτηση γιατί Κάποιες παρατηρήσεις που κάνατε με έκαναν να σκεφτώ τον τρόπο που, που ίσως υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στο κομμάτι της διακυβέρνησης και στο κομμάτι της ανάθεσης των καθηκόντων. Με την έννοια ότι εάν βγάλουμε το ενιαίο τον ενιαίο κανονισμό που συμφωνώ ε, δεν είναι αυτό το πιο επίμαχο ιδιαίτερα όμως όσον αφορά την σύγκληση της εποπτείας και την άμεση εποπτεία επίσης στον τομέα δηλαδή αυτών νομίζω πως το θέμα είναι του κατά πόσο στη διακυβέρνηση είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την συλλογική ιδιοκτησία γιατί δεν έχουμε τις εθνικές εποπτικές αρχές και την ΕΣΜΑ Έχουμε ε, την ΕΣΜΑ όπου οι επόπτες ε, συγκεντρώνονται και ίσως εκεί η διακυβέρνηση με κάποια ρύθμιση όπως είπε και ο Ζακ Τελαροζιέ εκεί να μπορούσε να υπάρχει περισσότερη ιδιοποίηση, ιδιοκτησία της, της υπόθεσης αυτής, γιατί εκεί σχηματίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εποπτεία. Όσο λιγότερο λοιπόν βλέπουμε αυτό το πρόβλημα, και υπερβολική αντίσταση, να λένε δηλαδή οι άλλοι, ναι, εγώ κάνω τι, δουλειά μου, τι, τι θέλουν τώρα αυτοί. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μία αγορά, κάποιοι να κάνουν τη δουλειά τους, είναι ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγορά. Πώς μπορούμε λοιπόν να δράσουμε πιο συλλογικά. Δεν λειτουργούμε σε ένα τέλειο κόσμο. Τι θέλει τώρα και η Επιτροπή, τι έρχεται και μας ζητάει. Εμείς τόσο καλά τα καταφέρνουμε. Ναι, το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα του να γίνουμε μία ενιαία αγορά, ιδιαίτερα όσον αφορά τι κεφαλαγορέ. Γιατί ο τραπεζικό τομέα είναι διαφορετικό. Εκεί συμφωνούμε με την κατανομή. Υπάρχει ΑΙΟΠΑ, άλλο ενιαίο, είχε, ε, ε, ενιαίο σύνολο κανόνα. περιπτώσει. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να συμφωνήσουμε με τρόπο ώστε να είμαστε αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τους ε, συμμετέχοντες στην ε- ε- ΕΖΑ. Μιλάμε για αναλογικότητα, για επικορικότητα, ότι πρέπει δηλαδή να γίνεται η άμεση υποπτία όταν χρειάζεται και να χρησιμοποιήσουμε την σύγκληση όχι ως επόπτη των εποπτών, αλλά ως μια, ένα κοινό τρόπο να έχουμε μια συνεπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ολόκληρη την Ένωση την Αυτή ήταν η ερώτησή μου και τώρα θα σας ζητήσω ακόμα και αν είχατε πολλές ε, και πλούσιες ερωτήσεις να μείνετε στα τρία λεπτά έκαστος για τα τελευταία, τις τελευταίες σας απαντήσεις. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος και θα εστιάσω στα, ε, στην περιπλοκότητα και το επίπεδο 1. Για να είμαι σαφής. Τι, θα μπορούσαν να κάνουν οι, οι συνομοθέτες, να διευκρινίσουν τα, τα ε, καθήκοντα στο επίπεδο 3, να τα πούν πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να μην δώσουν τις λεπτομέρειες στο επίπεδο 1, αλλά να διευκρινίσουν ε, τι πρέπει να, γίνει από, να κάνουν οι ΕΖΑ. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την αρχή της αναλογικότητας. Το δεύτερον, ε, γιατί παρατηρείται τόση περιπλοκότητα. Μπορούμε, μπορεί αυτό να αποδοθεί στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή από τις αγορές έχουμε έξι επίπεδα νομοθεσίας και είναι πάρα πολύ, είναι υπερβολικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρία επίπεδα και στο εθνικό επίπεδο άλλα τρία. <laughs> Είναι το τομείς ε, όπου χρειαζόμαστε περισσότερες κατευθύνσεις, ε, εκεί το αναλαμβάνουν τα Υπουργεία Είναι υπερβολικά όλα αυτά. Και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα καταλήξουμε σε, ένα πραγματικ... σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ώστε ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε να είναι 10-15 χρόνια, να έχουμε έναν κώδικα που θα αποτελείται από την νομοθεσία για τις κεφαλαγορές για όλα τα κράτη-μέλη. Σε ένα επίπεδο ώστε να μειωθεί ο περίπλοκος αυτός χαρακτήρας. Δεύτερο θέμα που είναι ένα Ηράκλειο έργο και δεν μπορώ να πω πώς ακριβώς θα γίνει. Ίσως αν αλλάξουμε τη διακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει το πράγμα. Να έχουμε δηλαδή ίσως περισσότερες αρμοδιότητες, να επιταχυνθεί η δραστηριότητα, Πάντως ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να επιτρέψουμε την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών. Υπό την αιγίδα των ΕΖΑ. Εδώ λοιπόν η αλλαγή πρακτικών είναι σημαντική. Δεν χρειάζεται δέ και καλά νομοθεσία. Να δούμε όμως πρώτα πώς θα λειτουργήσει η MIFID 2 και να έχουμε υπόψη ότι η προστασία του καταναλωτή δεν εξασφαλίζεται μόνο από την διοικητική νομοθεσία αλλά και από την ιδιωτική νομοθεσία και εδώ βλέπουμε να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στην Ευρώπη. Ο καταναλωτής ρωτάει, ναι, μπορώ να απαιτήσω ε, αποζημίωση, ναι ή όχι. Και ακόμα και εκεί πολλές φορές δεν είναι απλή απάντηση. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη εναρμόνιση και για την εντολή και τη... το κατά πόσον έχουν ξεπεράσει η ΕΖΑ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Εγώ ως καθηγητής νομικής μπορώ να πω μόνο πως σε κάποιες περιπτώσεις πολύ λίγες θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι, ξεπέρασαν τις αρμοδιότητες. Πάντως, ούτε η Κομισιόν, ούτε το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα ήθελαν να επεκταθούν σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Αυτά. Σχεδόν τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Yes, Κοιτάξτε. Κάτι επί της αρχής. Έχουμε δει διαφορετικές αντιλήψεις και συλλήψεις. Πρώτα απ' όλα η πρώτη, εν έχουμε ενιαίο επόπτη, αναφέρθηκε στο περίφημο Διοικητικό Συμβούλιο, συμβούλιο με πέντε προέδρους προετών. Μετά έχουμε το άλλο το συνεργατικό αυτό σχήμα, συνεταιριστικό δηλαδή μια οργάνωση που θα στηρίζεται στα μέλη. Πρέπει να βρούμε το μέσο όρο. Να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς πραγματικά ολοκληρωμένη εποπτεία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε έσμα, διότι ασχολούμαι με τις κεφαλαγορές και αναφέρομαι στο έσμα. Μία έσμα θέλουμε που είναι κάτι παραπάνω από μια ένωση, μια λέσχη εθνικών φορέων, NCAs. Θέλουμε να έχει πραγματική εξουσία συντονισμού, προώθηση εποπτική συγκλήσεω και να κατευθύνει τη δράση των εθνικών αρμοδίων αρχών. Προφανώς σεβόμενοι ότι η εποπτεία και εξουσίες βασίζονται στους εθνικούς φορείς. Είμαστε υπέρ σέσμα, Σημαντικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη της εποπτείας. Και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας πάντα το σχέδιο το τελικό που είναι η ενιαία κεφαλαγορά. Ευχαριστώ, Ανφιλή. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εποπτικών αρχών, δεν έχουμε αντίρρηση ο τομέας να πληρώνει μια εισφορά για τις εποπτικές δραστηριότητε. Αυτό ισχύει σε πολλούς άλλους τομείς. Και σε αυτό το τομέα έχουμε ζητήσει πολλά από τους φορολογούμενους. Θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των ελέγχων. Όσον αφορά την προστασία του καταναλωτού, πολλά μπορούμε να πούμε. Όλο και περισσότεροι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στις χρηματοστατικές υπηρεσίες υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς, η εφαρμογή των κανόνων επιτόπου αποκλίνει τεράστιες διαφορές από τη μία χώρα στην άλλη. Πώς να μιλήσουμε για ενιαία αγορά και να το συζητούμε αυτό συνεχώς χωρίς να φροντίσουμε για την πραγματική εφαρμογή ε, της νομοθεσίας επιτόπου. Να υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ένα consumer scoreboard όπου εκεί ταξινομεί τα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν οι καταναλωτές ε, βάσει διαφόρων κριτηρίων και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κάθε χρόνο έχουν τη χειρότερη θέση. Κάθε χρόνο τα ίδια. Το πρόβλημα της προστασίας του καταναλωτού δεν αφορά μόνο τις αποζημιώσεις, είναι σημαντικό αυτό και υπάρχουν, είναι κρίμα που δεν υπάρχουν και συλλογικέ δράσεις σε όλες τις χώρες. Χρειάζεται να κινηθούμε προληπτικά πολύ συχνά οι καταναλωτές και οι επαγγελματικοί χρήστες αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο προϊόντα περιπλοκότατα που δεν αντιστοιχούν σε ανάγκες τους και ε, μπαίνουν μέσα στη δίνη επιθετικών εμπορικών πρακτικών. Λοιπόν, είναι σαφές το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Οι εθνικοί φορείς, οι ΕΣΑΣ έχουν αρμοδιότητα εκεί αναφέρονται ότι οι εξουσίες που τους ανατίθενται σε θέματα εκδόσεως, ειδοποίηση, απαγόρευσης κάποιων προϊόντων, οι αρμοδιότητε δεν είναι σαφείς και γι' αυτό δεν έκαναν μεγάλη χρήση των καταλήλων μέτρων. Αυτό ισχύει, θα πρέπει λοιπόν να ξανά αναφερθούν οι αρμοδιότητε. Θα πρέπει η εντολή που θα δοθεί να είναι σαφή, επακριβή, θα αναφέρεται στον κανονισμό, τόσο ώστε να μην υπάρχουν πλέον δυνατότητε να αναφέρεται ότι εσά δεν έχουν ρόλο να παίξουν. Και γι' αυτό Είμαστε υπέρ ενός προϋπολογισμού για την προστασία των καταναλωτών στα πλαίσια των κανόνων των επιχειρηματικών και θα ανατίθενται στι τρει εποπτικέ αρχέ. Η ΔΕΜΗ δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι καταναλωτέ και οι χρήστε των χρηματοστικών υπηρεσιών είναι οι φτωχοί συγγενεί του χρηματοστικού τομέα. Και το άλλο. Χρειάζεται και το θέμα των βιωσίμων χρηματοστικών να μπουν μέσα στα πλαίσια της εποπτείας του τομέα. Ο Φελίξ Χούφελτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και να αναφέρω και εγώ κάποια ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι τέθησαν ως ερωτήματα προς εμένα. σας το θέμα του ότι ενθαρρύνω το νομοθέτη σε επίπεδο πρώτο επίπεδο να είναι πιο συγκεκριμένο. Όχι, αυτό είναι παρανόηση. Είναι η φύση του νομοθέτη να κάνουν πολιτικούς συμβιβασμού. Ό,τι και να σημαίνει αυτό εγώ, απλά προσπαθούσα να εξηγήσω. Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει πιο συγκεκριμένη νομοθεσία σε ρύθμιση μάλλον σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Γιατί σε επίπεδο Πρώτο επίπεδο, η νομοθεσία είναι διαφορετική στη φύση τη. Δεν θέλω να είμαι αφελή για την νομοθεσία πρώτο επίπεδου. Όχι. Όσο πιο πολύ ασχολούμαι με την ρύθμιση εγώ ίδιο, τόσο πιο πολύ ε, βασίζομαι σε αρχές και όχι σε νομοθεσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, απλά για να αποφύγω την παρανόηση αυτή. Δεύτερο σημείο. Ο κύριος ε, Κλίντ έκανε μια περίεργη ερώτηση, αστεία κάπως. Κατά πόσον μια εθνική αρχή ενδεχομένω να σαμποτάρει την νομοθεσία αν ε, περιλαμβάνει αρμοδιότητα, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκέ αρχές. Εμείς είμαστε δημόσιε αρχές. Δεν σαμποτάρουμε. Τους πολίτε εξυπηρετούμε. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μα. Άρα, δεν πιστεύω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Ένα προφανές παράδειγμα ήταν η δημιουργία της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Ε, είμαστε αναπόσπατο τμήμα της ε, και δουλεύουμε σκληρά για να πετύχει. Αλλά όπως είπα και εισαγωγικά. Άλλο είναι, πιστεύω, να συζητάμε ανοιχτά το ότι πιστεύουμε ότι αποτελεί καλή ευρωπαϊκή πολιτική ή όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να σαμποτάρουμε κανέναν. Διάφοροι βουλευτές είπαν για την Λετωνική Τράπεζα, την LBRV. Και μιας και συμμετέχω στη λήψη αποφάσεων, δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί μου απαγορεύεται. Αλλά βασικά η κατάσταση είναι η εξή. Πρόκειται για μία αρχή η οποία εξέφρασε ανησυχίες για περιστατικά για εξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε ό,τι αφορά την τράπεζα αυτή. Ξεκίνησε λοιπόν μια κρόαση επί 60 ημέρες. 60. Αυτό προφανώς και δημοσιεύτηκε ως γεγονός. Αυτό είναι αρκετά θετικό και καταδεικνύει πόσο ευαίσθητες είναι οι τραπεζικές καταστάσεις. Αυτό όμως επηρέασε την ρευστότητα της τράπεζας δραματικά. Μάλιστα. 70, σε 72 ώρες, ε, σε 3-4 μέρες. Και έτσι η τράπεζα έφτασε στο χείλος της αφαιρεγγιότητας. Και έτσι ο επόπτης μέσα σε λίγες ώρες αναγκάστηκε να λάβει δραστικά μέτρα. Ένα μνημόνιο, μία δήλωση αποτυχίας ή πιθανότητας αποτυχίας την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα ακριβώς αυτά κάναμε και αυτά συζητούσαμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια. Το θέμα ποιο είναι ότι οι δραστηριότητε για την αιμοποίηση παρανόμων εσόδων είναι αυστηρός σε εθνικό επίπεδο. Άρα υπάρχει μηδενική αρμοδιότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν λοιπόν και ο πυρήνας του, προβλέμ, του προβλήματος. Τα προβλήματα ρευστότητος, ε, αντίθετα με τα προβλήματα κεφαλαίου, μπορούν ε, να παρουσιάσουν προβλήματα μέσα σε λίγες ώρες. Άρα, αν αναζητάτε εγγυήσει ε, για το κατά πόσο αυτό θα ξανασυμβεί στο μέλλον, η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Και οι επόπτες έχουν καθήκον να διαχειριστούν τι συνέπειε. Αν όλοι πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητε για την ομιμοποίηση παράνομων εισόδων. Από ό,τι ξέρετε το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, μην σα πω και παγκόσμιο. Αλλά η εποπτεία είναι σε εθνικό επίπεδο, αυστηρά. Αν αλλάξει αυτό, φυσικά θα χρειαστεί πολιτική συζήτηση. Πολιτική συζήτηση την οποία εγώ δεν μπορώ να αλλάξω με το ρόλο μου. Είναι ευρύτατη η πολιτική συζήτηση. Αν δεν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, εξαρτώμαστε από τις εθνικές αρχές, από τις λιτονικές αρχές στην προκειμένη περίπτωση. Αυτά για τη Λιτωνική Τράπεζα. Δύο σύντομες τώρα απαντήσει επιτρέψτε μου, για την κοινή κουλτούρα των εποπτών. Αναφέρθηκε επανελειμμένα και όντω, αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά πλέον εκτήματα των δομών μα. Εγώ να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία το εξής. Ο τρόπος ε, με τον οποίο δρούν και αντιδρούν οι επόπτες και δρούν ανάμεσα τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφέρει ολοσχερό σε σχέση με αυτό που γινόταν πριν από 10-15 χρόνια. Αυτή η διαρκής ε, διάδραση, αυτή η ε, διαρκής ροή ε, πληροφοριών έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είμαστε σε τέλειο επίπεδο, αλλά έχουν αλλάξει πολλά. Να πω και κάτι άλλο. Το οποίο το είπαμε και προηγουμένω και ισχύει όχι μόνο για την προστασία των καταναλωτών, αλλά γενικώ πώ, θα ήταν λάθο να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και ίση αντιμεταχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο μέσω του χρηματοοικονομικού κανονισμού. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί νομικοί τομεί ε, που δεν έχουν αρμονιστεί καθόλου. Αφαιρεγγιότητα, πρόσβαση στα δικαστήρια, ε, αστικό δίκαιο και αν θέλουμε δηλαδή να τα περάσουμε όλα μέσα από τον χρηματονομικό κανονισμό, θα αποτύχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποτίμηση των πόρων που χρειάζονται, σε περίπτωση που όλα αυτά μεταφραστούν στην πράξη, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή υλοποιηθεί, εγώ προσωπικά τι πιστεύω, ότι οι πόροι που διατίθενται, περίπου 200, είναι υπερβολικά χαμηλοί με μεγάλη διαφορά από την εμπειρία μου στην τραπεζική εποπτεία. Εγώ θα ήθελα να τριπλασιαστούν, να τετραπλησιαστούν. Μη σα πω και ότι αυτό θα προωθηθεί και στι εθνικέ αρχές, ούτε και θα λάβουμε του ε, πόρους μας. Αυτό όμως είναι το δευτερεύον πρόβλημα. Το βασικό θα ήταν να σκεφτούμε και κάποια από τα βασικά στοιχεία ε, ε, επί τη αρχή. Ευχαριστώ, λέει και ο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος. Έχετε δίκιο. Όταν προσπαθήσαμε με την οδηγία να εισαγάγουμε κάποια στοιχεία για την υποπτική σύγκληση, αντιμετωπίσαμε τείχος, τείχος από πλευρά του Συμβουλίου στους τριμερείς διαλόγους. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ο κ. Τέλα Ροζιέρ. Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε αργήσει. Ε, I think you raised a very... Προς την κύριε μπορώ να πω ότι πιστεύω πως αναφέρατε ένα πολύ καλό ερώτημα για την εποπτεία. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας για την εποπτεία των, ε, ε, των CSD ή των ICSD. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε αν αυτά είναι συστημικά, όπως και τα CCP ένα ανοιχτό το ερώτημα. Και η Γκόλντα ESRB. Γιατί είναι η ESRB. Πιστεύω πως κάτι νομίζω ότι θα, θα πρέπει να είναι μικρότερο από ότι σήμερα. Θα πρέπει να αποσπαστεί από το ECD. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα ήταν σκόπιμο λόγω των συνηθιών που έχουν ε, καθιερωθεί στη διάρκεια των ετών. Θα νομίζω πως θα ήταν καλό θα πρέπει να είναι υπόλογοι για το τι προτείνουν και τι λένε. Ζούμε πάντως σε περίπλοκο και επικίνδυνο διεθνές σύστημα και δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η SRB που είναι τελείως συνδεδεμένη με, μια από τις με τους μεγαλύτερους φορείς ε, στην, ε, στο διεθνές προσκήνιο έχει την ε, ανεξαρτησία και την ποιότητα Άρα λοιπόν το θέμα είναι τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Θέλουμε να έχουμε έναν ναύτη πάνω πάνω στο κατάρτι και να είναι υπεύθυνο για τις παρατηρήσεις που κάνει, για τις προειδοποιήσεις που δίνει, για τους κινδύνους, τους πιθα... τα πιθανά αίτια ρήξης ή διακοπής. More specifically to Mr. Giegold, who said, you know, you're all speaking of το γεγονός ότι αυτή η εποπτεία δεν ε, εφαρμόζεται με εναρμονισμένο τρόπο. Τι να σας πω. Ναι, λέμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ισότιμο πεδίο, να, είμαστε, να έχουμε ισχυρή υποπτική σύγκληση. Μα δεν κάνουμε έτσι τίποτα όμως. Έχω μια-δύο προτάσεις. Πρώτη πρόταση. Να χρησιμοποιήσουμε ε, και να πούμε ότι είναι σχεδόν προφανής η υπόθεση της μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Νομίζω ότι είναι αυτό πολύ σημαντικό, δεν είναι απλά μια δυνατότητα, μια πιθανότητα μάλλον, είναι κάτι, για, για τους ανθρώπους που είναι δυσαρεστημένοι, είναι κάτι το οποίο θα επιβληθεί από την εκάστοτε ε, εποπτική αρχή. Θα έλεγα λοιπόν πως η εποπτική αρχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ξεκινάει ε, να, μια διαδικασία δια, ε, διατησίας. Γιατί αυτό μας δίνει μια αίσθηση ευθύνης όταν υπάρχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας. Το δεύτερο είναι ότι αν παρά την διατησία που ξέρουμε ότι δεν είναι πάντοτε άμεσα επιβλητέα μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας, αν λοιπόν παρά την διατησία το πρόβλημα της μη εφαρμογής παραμένει, τότε οφείλει η ΕΣΜΑ ή και άλλοι, είπα την ΕΣΜΑ γιατί φροηδικά ε, ολίθισα Πάντως ε, είναι, ε, είναι ευθύνη των αρχών να ζητήσουν από το δικαστήριο να συμβουλέψει κάθε φορά και να το κάνει αυτό με, σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, προθεσμίες. Γιατί αυτές είναι οι μικρές μου προτάσεις προς τον κύριο Γκόλντ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ζητήσω από τους συνεισηγητές να συνοψίσουν πολύ πολύ σύντομα, γιατί βεβαίως δεν πρόκειται για το τέλος της συζήτησης σήμερα. Παρακαλώ. Ο κ. Μπάλτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και όλους τους πανελίστες για μια φορά ακόμα. Να πω ότι έχω και κάποιες θετικές παρατηρήσεις ε, σε σχέση με, σημερινές, ε, με τη σημερινή συζήτηση και να πω ότι άκουσα και, και ευρία κριτική κατά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με την κριτική αφενός κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι κι εγώ ίδιος πόση δουλειά, πόση δουλειά και εγώ και η κυρία Περές ε, θα έχουμε και φυσικά και οι υπόλοιπε κοιόδες εισηγητές. Τεράστιος όγκος δουλειάς για να επεξεργαστούμε τις προτάσεις αυτές. Αυτό που συγκρατώ από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει οριστική ακόμα ε, τοποθέτηση. Η αναλογικότητα δεν είναι μόνο θέμα ε, νομοθεσίας πρώτου επίπεδου, αλλά και δευτέρου και τρίτου επίπεδου. Οι αποπτικές αρχές επίσης ε, χρειάζονται πιο πολλές κατευθυντήριες γραμμές για αναλογικότητα, για να δρουν, και να διοικούν. Και σήμερα λοιπόν προτάθηκε η αρχή της αναλογικότητας να εφαρμοστεί και να κατοχυρωθεί και στον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και οι υπόλοιπε μελέτες θα πρέπει να κάνουν τη σύνδεση με το στοιχείο αυτό. Κάτι άλλο που είναι σαφές επίσης, ε, ότι χρειάζεται καλύτερη διάκριση μεταξύ ε, ρύθμισης και εποπτείας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό για τη σύνθεση και τη χρηματοδότηση των αρχών. Τρίτο στοιχείο. Οι άμεσες αρμοδιότητες της ε, ΕΣΜΑ φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται με κριτικό πνεύμα συνολικά και επίσης ό,τι αφορά την εποπτεία των σε θα πρέπει να δούμε στη σχετική νομοθεσία τι θα γίνει και φαίνεται ότι η πιο πολύ είναι διστακτική σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των άμεσων αρμοδιοτήτων της ΕΣΜΑ για τις ε, Γρήγορε αλλαγέ Αυτό και εγώ το σύμφωνο, με αυτό δεν την χάνουν υποστήριξη. Χρειάζεται ρεαλιστική και πραγματιστική προσέγγιση για το ποιε είναι, ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία ήδη έχουν αναλάβει ή μπορούν να λάβουν στο μέλλον οι εθνικές αρχές, στο θέμα των τρίτων κρατών τώρα. Και εδώ θα έχουμε πολλά να κάνουμε και θα πρέπει σίγουρα στην έκθεσή μας να κάνουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο την προδιαγραφή των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών για το μοντέλο διακυβέρνηση, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Τι ακούσαμε με σαφήνεια, ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε πιο πολύ προς την κατεύθυνση της λιγότερης πολυπλοκότητας και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. και θα πρέπει να κοιτάξουμε και τι γίνεται με τους εμπλεκόμενους φορεί σε κάθε περίπτωση. Α, κάτι άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον, η παρατηρήση του κ. Ντουλαροζιέρη για την ε, ενίσχυση της ανεξαρτησίας ε, της Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και την αποσύνδεση από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σε σχέση με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Τέλος, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση εισακούσαμε τις ε, προτάσεις και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων σήμερα το πρωί και σίγουρα θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερο στην κατάρτιση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ Περβάνος Περές, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας. Επειδή τους έχουμε σαν επιλεγμένους συνεισηγητές, αυτό δεν σημαίνει συμφωνώ μαζί τους, αλλά ήταν πολύ καλή λύση που διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη θητεία, ποιοτική συμμετοχή των παρισταμένων. Και σας ευχαριστούμε. Δώσατε κάποια στοιχεία σημαντικά. Το θέμα είναι δυσχερές υπάρχουν και αντικρουόμενε ζώνες στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο. Το πεδίο αρμοδιοτήτων Φερρυπίν, η διακυβέρνηση και η χρηματοδότηση. Σε κάθε μία πτυχή μας διαφωτίσατε, μας δώσατε ιδέες. Η συνεισφορά σα. είμαι σίγουρη ότι θα συμβάλλει στην τροφοδότηση του προβληματισμού μας και θα καταλήξουμε συγκεκριμένε προτάσει. Συγκρατώ σε βασικό μήνυμα το θέμα του χρόνου. Και αυτά που είπε ο Βολφ Κλίντς, ο σκιώδης ηγητής των φιλελευθέρων. Αυτή η επανεξέταση του θέματος ΝΕΖΑ πρέπει να τελειώσουμε και τη θητεία, συμφωνούμε. Ελπίζουμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον και να μην θεωρήσουμε ότι αυτή η αναθεώρηση μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και θα κάνει νέα αναθεώρηση, νέα θητεία των ΕΣΑ. Πρέπει να είμαστε μελλοντοστραφείς και να δώσουμε τα κατάλληλα μέσα σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς φορείς ελέγχου. Όσον αφορά το ECRB, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε στοιχεία πολύ light όσον αφορά τις αλλαγές. Και ίσως χρειάζονται τα μέσα να εξετάσουν περαιτέρω τις αρχές, τις αρμοδιότητες. Και όπως είπε και ο Ντελαροζιέρ, θα πρέπει το CRB να γίνει πραγματική ηθική αρχή, αν θέλετε, εντολογική αρχή. Κατανοώ την ιδέα που διέπνευσε την έκθεσή σας. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη μακροοικονομικής εποπτείας. Ικανοποιητικό διανοητικά. Σήμερα όμως δεν μπορούμε πλέον στο παρόν πλαίσιο να ονειρευόμαστε. Δεν ξέρω ποιον το αντίστοιχο αυτής αρχής της είπα, ΕΕ, αν υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η πτυχή. Παράλληλα με την εφαρμογή ε, της, ε, ενιαίας, ε, της υλοποίησης ενιαίας κεφαλαγοράς. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στις αρχές των CDS, αν είναι συστημικό μέσο ή όχι. Ίσως πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο την κατάσταση με μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη. Άκουσα πολλές παρεμβάσεις που ήταν χρήσιμες. Αφορούσαν τη σχέση μεταξύ αρμοδιοτήτων και ρόλου των ΕΣΑ και του δικαστικού συστήματος. Η σχέση με το δικαστήριο. Σε άλλους τομείς έχουμε την εντύπωση και την ιδέα όσον αφορά τη λειτουργία των χρηματοστατικών αγορών, η προσφυγή στο δικαστήριο δεν συμβαίνει αρκετά συχνά ή τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Συγκρατώ και άλλα τρία σημεία. Το πρώτο. Αυτό που τονίζεται στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τονιστεί περαιτέρω, δηλαδή διαφοροποίηση όσον αφορά τη λειτουργία και το ρόλο και τη σχέση με τους τρεις φορείς, μεταξύ των τριών φορέων. Δεύτερον, στο θέμα των καταναλωτών. Εκεί προφανώς πρέπει να προσπαθήσουμε σαν Ευρωκοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε την πρόοδο του τομέα για τη διακυβέρνηση. Μάλλον σύγκληση, όχι διακυβέρνηση, σύγκληση, διορθώνει η ομιλήτρια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε εκτός τον έλεγχο ομοτήμων αλλά ίσως βάσει της προτάσεως του Ευρωκοινοβουλίου του 2014 να έχουμε ένα δίκτυο επιδόσεων, ένα scoreboard, σύστημα βαθμολόγησης, ένας ρυθμός προόδου που πρέπει να συγκρατηθεί και να είναι προτεραιότητα αυτό για μας. Σας συνεισφορά το Ευρωκοινοβούλιο αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θεωρώ ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες ακροάσεις μας. Χρησιμότατη. Ευχαριστώ τους διατεκριμένους, προσκεκλημένους μας, Ρούντι Γκερβάλλα, Σεβαστιάν Αρμπέλα, Ανθιλή, Φέλιξ Χούφελτ και Ζακ Ντελαγοζιέρ, Σας ευχαριστώ. Σημαντικότατη συνεισφορά σας. Το χρονοδιάγραμμα, όπως ξέρετε, είναι ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Αλλά υφίσταται. Παρουσίαση σχεδίου εκθέσεως 18-19 Ιουνίου, ημερομηνία τροπολογία 9 Ιουλίου, εξέταση τροπολογιών 3 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 24 Σεπτεμβρίου. Έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε τιμέ διαλόγου τον Οκτώβριο. Για να ολοκληρωθεί το θέμα εγκαίρως, πριν το τέλος της θητείας. Θα πρέπει να τηρήσουμε, πιστεύω, αυτό το χρονοδιάγραμμα και να προσπαθήσουμε να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία στη θητεία μας ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά την σύνταξη των άρθρων, να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ. Και πάμε σε κάποιο παράπλευρο αποτέλεσμα της αναθεωρήσεως. Καθίστε εκεί, είσαστε εισηγητής. Λοιπόν, κερδίζω χρόνο για να παρουσιάσω το νέο θέμα, το επόμενο. Το παίρνουν την εθόρυση των ΕΖΑ, αλλά πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί πιο σύντομα. Αφορά την έδρα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών μάλλον. Σας έδωσα κάποιο χρόνο, περισσότερο έδωσα χρόνο στην ακρόαση, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και ψηφοφορία. Έχουμε δύο σημεία. Σας ευχαριστώ εκ νέου, ευχαριστώ εκ νέου όλους τους ομιλητές μας. Ως γνωρίζετε λοιπόν, ένα από τα στοιχεία προς εξέταση είναι η έδρα. Από πλευρά Συμβουλίου ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία, κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα το Συμβούλιο, δεν είναι μόνο θέμα περιεχομένου, Η θέση του εισηγητού συμπίπτει με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τίθεται θέμα διαδικαστικό όμως και θεσμικό. Οπότε το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκαθαρίσει το ότι η συναπόφαση είναι συναπόφαση. Η συναπόφαση είναι μια διαδικασία. Οι, δύο συνομοθέτες συναποφασίζουν. Τι σημαίνει αυτό ότι έχουν τη δική τους εξουσία, είναι κυρίαρχοι φορείς. Ή οδήποτε άλλο στοιχείο ε, είναι υποδέστερο, διότι έχει κυριαρχία το σώμα αυτό. Είναι καλό το ότι σε αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο προτείνει το ίδιο, καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα όπως και το Συμβούλιο. Αλλά είναι χρήσιμο ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι κινείται στα πλαίσια της κυριαρχίας του και δεν έχει νομικούς δεσμούς και περιορισμούς από οποιαδήποτε διαδικασία που βέβαια δεν είναι και τέλεια διαδικασία αξιολογήσεως και εγώ συμφωνώ με τις επικρίσεις που αναφέρονται στην έκθεση περί της διαδικασίας αλλά αρκετά είπα ο Μπούρχα το εισηγητής Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αναφέρατε με το σχέδιο έκθεσης. Άσκουμε ε, σαφή κριτική και τα προβλήματα που έχουμε σε ό,τι αφορά την ε, λήψη αποφάσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ως συνομοθέτης έχουμε ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της έδρας. Ίσο δικαίωμα με αυτό του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν η λήψη αποφάσεων και το 2010 ήταν σαφές τότε για η ΟΠΑ, η ΕΣΜΑ και η ΕΜΠΑ αποφασίστηκαν από την Επιτροπή, το Συμβουλίο και την Κοινοβούλιο. Ήταν μια διαθεσμική συμφωνία τότε. Είχαν γίνει τριμερείς διάλογοι, διαπραγματεύσεις και ως εκ τούτου ζητούμε από το Συμβούλιο περαιτέρω πληροφορίες για το πώς κατέληξε στη λήψη αποφάσεων και κυρίως τα κριτήρια, πώς τα ζήγησε για τη συναπόφασή μας λοιπόν. Δεν μπορεί. Είχε γίνει μια κοινή δήλωση το 2012, αλλά η κοινή δήλωση δεν είναι κανονισμός. Ούτε μια κοινή δήλωση μπορεί να αναιρέσει την συναπόφαση και η κοινή δήλωση από την οποία λείπει η άποψη του Κοινοβουλίου δεν είναι πλήρης, πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε έγκαιρη μεταρρύθμιση αναθεώρηση τη κοινή δήλωση και ακριβώ αυτό λείπει. Μία διαφανή διαδικασία. Έγκαιρη ίση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη και να εγγυάται αυτό και παράλληλα τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων να ε, έχουν ίση πρόθεση. Άρα θεωρούμε, καταρχάς να θυμηθυμίσουμε ότι είναι τρεις διαφορετικές αυτές οι υποπτικές αρχές και οι οι οικονομικές αρχές ε, χρειάζονται και την εμπειρογνωμοσύνη και την εποπτεία. Αυτό διαφαίνεται και σε διεθνές επίπεδο, στον τραπεζικό κλάδο, στα αξιόγραφα, στις ε, ασφάλειες. Όλα αυτά διακρίνονται. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων, η Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχουν διαμορφωθεί προς, και έχουν εξελιχθεί προς διαφορετική κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την οργάνωση τους. Θα ήθελαμε να επιβεβαιώσουμε ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα, οι αρχές αυτές από γεωγραφική άποψης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η Περβάνος στο ίδιο πνεύμα με τον κύριο Μπάλτς από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Του τουλαχθέντος. Αυτό μου θυμίζει επίσης αυτό που έγιναν και στην τελευταία διαπραγματεύση για το που Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είχε παρουσιάσει προτάσεις οι οποίες εξαρτώνταν από τον συνομοθέτη ουσιαστικά όμως. Στο Συμβούλιο έχει αυτή την κακή συνήθεια. Είναι 27 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και θεωρούν ότι μπορούν να πούν στους νομοθέτες τι να κάνουν. Μα δεν γίνονται έτσι όμως τα πράγματα και προφανώς και μας ακνευρίζουν γιατί αν μπορεί να γίνει αυτό για ένα θέμα μπορεί να γίνει για όλα του τουλεχθέντος. Υπάρχουν νομίζω διάφορα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Καταρχάς, ότι ο συνεισηγητής ε, δεν αμφισβητεί την ουσία της ε, απόφασης. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή στην ίδια κατάσταση που βρισκόμασταν και για τα άλλες αρχές για τον Brexit. Απλά θέλουμε να υπάρχουν οι βέλτιστοι όροι. Αποφασίσαμε λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι. Αν η Ευρωπαϊκή Τραπεζική αρχών μπορεί να εγκατασταθεί στο Παρίσι πρωτού γίνει το Brexit, πριν το Μάρτιο του 2019 δηλαδή. Θέλουμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Θέλουμε εγγυήσει. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να εισακούσει το Συμβούλιο. Θέλουμε να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για την κοινή δήλωση, η οποία προφανώς έχει εμπνεύσει τις εργασίες του Συμβουλίου, αλλά δεν έχει οδηγήσει σε μια καλή μεθοδολογία, βρίσκουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε από τον συνεισηγητή και επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Το θέμα του συγκεκριμένου χαρακτήρα των αρχών θα πρέπει να γνωρίσουμε και στο πλαίσιο της κοινή δήλωση και των τροπολογιών τις οποίες ακόμα συζητιούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής ε, προπολογισμού. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν ε, συνεργίες ε, στους ε, σωστούς τομείς, σε θέματα υπηρεσιών, σε θέματα αρμοδιοτήτων, γιατί αν υπάρχουν διάφορες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πόλη, προφανώς υπάρχουν και συνέργειες σε ό,τι αφορά το υποστηρικτικό σκέλος και να υπογραμμίσω τέλος την άποψη την οποία ανέκρινε η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων χθε και περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις που θα μπορέσουν να προταθούν. Φυσικά, αφότου εμ, καθαρίσουμε το κείμενο από διάφορες ασάφειες τις οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και όντω θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή ε, στις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ πόλει, το Συμβούλιο ανέφερε ότι κακώ απευθύνονται αυτέ οι εκκλήσει ε, στο Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι το Συμβούλιο αυτό που λαμβάνει τι αποφάσει και ήταν συμφωνίες πολιτικές εκτός του κόλπου του Κήτου Συμβουλίου. Άρα νομικός πως τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να υπερψηφίσουν κάτι στον τρέμερη διάλογο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι νομική διαδικασία. Τα υπόλοιπα δεν έχουν νομική υπόσταση. Και νομίζω ότι καλά κάνουν οι συγητές και μας το υπενθυμίζουν. Η κυρία Σφίνμπορν. Σα ευχαριστώ. Και αυτέ δεν είναι δικέ μου απόψεις, είναι του σκιώδου που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και μου ζήτησε να διαβάσω ένα σύντομο, μια σύντομη δήλωση όσοι δεν είστε. Συμφωνεί με την πρόταση, αλλά και με τι πρότασίε ένα και 2 των συνεισηγητών. επίση εκτιμά το, το στόχο τη τροπολογία 4 των συνεισηγητών, μια εκδοχή τη οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κανονισμό EBA κύριος Λούνε συμφωνεί ότι η τοποθεσία θα πρέπει να επιλεγεί μέσω μιας διαφανής, διαφανούς διαδικασίας και αναγνωρίζει ότι θα μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία. Θα σκέφτεται περισσότερο για τη συγκεκριμένη διατύπωση της τροπολογίας αυτής και των ε, αιτιολογικών σκέψεων. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κλίντς έφυγε. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές, την Περβάν Μπερές και τον Μπούκχαρτ Βάλτς, για το σχέδιο που μας έστειλαν. Και θα ήθελα να επικρίνω και εγώ έντονα, όπως έκαναν ήδη οι δύο συνεισηγητές, τον τρόπο που λήφθηκε η απόφαση αποκλειστικά από το Συμβούλιο, χωρίς την απαραίτητη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου τόσο στον ορισμό των κριτηρίων, όσο και στην απόφαση για τη νέα έδρα όπως θα έπρεπε, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Αυτή η μέθοδος λήψης αποφάσεων είναι απαράδεκτη, παρά το γεγονός ότι δεν έχω αντίρρηση με την επιλογή του Παρισιού. Πιστεύω ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε υποστηρίζοντας τη δημοκρατική λογοδοσία, τη διαφάνεια, τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Η ομάδα μου, όπως γνωρίζετε, έχει εκφράσει ενστάσεις και στο παρελθόν για το ρόλο αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όπως και για το γενικότερο σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Τούτη την ώρα όμως νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην υπεράσπιση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου ως συνομοθέτη και να προκαλέσουμε με αφορμή και, ε, αφορμή και αυτό το θέμα μια ουσιαστική συζήτηση με το Συμβούλιο για το πώς θα εφαρμοστούν όσα έχουν αποφασιστεί και ισχύουν ήδη από το 2012 που ενισχύουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη των αποφάσεων και επομένως και των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την ίδια την αρχή, την Ευρωπαϊκή των Τραπεζών, νομίζω ότι έχει σημασία μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική μετεγκατάσταση και έγκαιρη και κριτήρια που να εξασφαλίζουν και τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους και με αφορμή αυτό να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εύρυθμη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Αρχών και της συγκεκριμένη Αρχής Τραπεζών. Επιφυλάσσομαι στη διάρκεια της υποβολής των τροπολογιών και της σχετικής συζήτησης να συνδράμω σε αυτό το πνεύμα τους δύο συνεισηγητές. Ευχαριστώ. Uh, Molly, are you speaking on behalf of Sven Giegel? Molly, θα μιλήσεις εξ ονόματος του Σβέν. Ναι, αλλά για την Ευρωβινιέτ. Άλλος σκιώδης δεν βλέπω. Catch the eye. Hayes. Um, president, as, as, uh... Πρόεδρε, εγώ είμαι MP. Είμαι προβουλευτής από τη χώρα που έχασε όταν uh, έγινε η κλήρωση για την Eurovision και θέλω να υποβάλω το, να πω μάλλον ότι ο τελείως αδιαφανής τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτος. Το πιο σημαντικό είναι τώρα να υπάρξει βεβαιότητα όσον αφορά το προσωπικό της ε, τραπεζικής αρχής αφού θα μετακινηθεί στο Παρίσι. Βέβαια, σωστό είναι να πούμε ότι ναι, είναι καλύτερο από άποψη εξοικονομήσεων για να έχουμε δύο οργανισμούς στην ίδια πόλη. Όμω είναι επικίνδυνο προηγούμενο. Δύο οργανισμοί να είναι στην ίδια πόλη. Λάθος μηνύματα στέλνει στην Ευρώπη, στις μικρότερε χώρες, στι περιφερειακές ε, ε χώρες. Ε, δεν είναι καλή αρχή. Και ξέρω ότι γίνεται λόγω της διαδικασία, αλλά μια λύση μακροπρόθεσμα θα ήταν ίσως να μην στείλουμε αυτά τα λάθος μηνύματα. Όταν ε, η Κομισιόν λοιπόν εξετάζει όλες τις προσφορές, καλό θα ήταν να γίνεται να, δημοσίευση της θέσης και της αξιολόγησης της Κομισιόν. Άρχεται η Κομισιόν εδώ στο Κοινοβούλιο να ρωτάμε ερωτήσεις. Αυτός είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε τις συμφωνίες ε, που γίνονται ε, στα κρυφά. Πάντως ε, συμφωνώ με τους συγητές, έχουν πει σωστά τις αρχές για την αναθεώρηση, τα σωστά κριτήρια αλλά ε, το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε και να δώσουμε βεβαιότητα τώρα στο προσωπικό τη CBA και στην ίδια την αρχή, καθώς θα μετακινηθεί στο Παρίσι. Καλή επιτυχία λοιπόν για το μέλλον. Thank you. Marcus Ferber. Ευχαριστώ κύριε Σφέρμπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μικρή παρατήρηση μετά την ε, έκθεση χωρίς απαλλαγή που ήμουν υπεύθυνο του περασμένο έτος και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε διάφορες συνεργίες στις αρμοδιότητες. Τότε λοιπόν ε, μια ομάδα πολιτική ε, μαζικά με επέκρινε και τελικά δεν πέρασε αυτή η απόφαση μου. Κάνει λοιπόν εντύπωση ότι αυτοί που πέρσι ασκούσαν κρατική τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Σωστό ήταν ή λάθος ο Πρόεδρος να χρησιμοποιήσουμε και τη διαδικασία Catch the Eye, γιατί αυτό που επικρίθηκε τότε δεν ήταν το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να συναποφασίζει, αλλά το ότι θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, όχι στη χορήγηση απλαγής. Υπάρχουν δύο τρόποι, θεωρώ. Είτε το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει από την αρχή, είτε το Κοινοβούλιο δεν θα δεσμεύεται από αυτά που αποφασίζει το Συμβούλιο. Δεν γίνεται όμως και τα δύο, ούτε να έχουμε συμμετοχή, αλλά να είμαστε πολιτικά και ηθικά υπεύθυνοι. Νομίζω ότι καλά θα κάναμε να το διευκρινίσουμε το θέμα αυτό και να ασκήσουμε κριτική. Η η, πολιτική του νύπτου του Συμβουλίου. σε ό,τι αφορά δηλαδή τον εντοπισμό των κριτηρίων, των δικαίων λύσεων και να μην είμαστε υπεύθυνοι για τίποτα σε τελική ανάλυση. Είπαμε ότι ναι, Μπορεί να υπάρχει ισοψηφία. Ισοψηφία βέβαια με 27 δεν θα υπάρχει, αλλά μπορεί κάποιος να απόσχει. Δεν ξέρουμε. Ειλικρινά θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες του πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα η Ευρώπη. Δεν αμφισβητούμε το περιεχόμενο λοιπόν, να το τονίσουμε αυτό. Από θεσμικής και πολιτικής άποψης έχουμε αντιρρήσεις. Οι η κυρία Περέζ. Ε, ε, l'importance de rassurer euh, le personnel des débat et la continuité de l'agence parce que je crois que ça doit être euh, notre fil conducteur. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε την σωστή προσέγγιση. Όσον αφορά τα λοιπά, το Συμβούλιο ελπίζουμε ότι θα απαντήσει με λογικό τρόπο στο αίτημά μας να ξανανοίξει το εκείνη δήλωση Ελπίζω να κάνουμε μια θεωρητική προσέγγιση, διότι ελπίζουμε τις επόμενες δεκαετίες να μην πρέπει να μεταγκαταστήσουμε μια υπηρεσία λόγω αποχωρήσεως ε, ενός κάτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Ο αντιπρόεδρος αναφέρθηκε σε κάποια αντίθεση που ίσως προκύπτει από αυτό που ζήτησαν να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των φορέων που εδρεύουν στο Παρίσι. Η συζήτηση ήταν ζωηρή τότε που είχαμε γνωμοτήσει του προπολογισμού και βασιζόταν επί των κριτηρίων που θα πρέπει να διέπουν την απόφαση για την έδρα των υπηρεσιών. Και το μόνο κριτήριο που ο τότε συγκριτής θα συγκρατήσει ήταν το κριτήριο ε, των ενοικίων των 10 υπηρεσιών. Και στην κοινή δήλωση το Ευρωκοινοβούλιο δεσμεύτηκε να ακολουθήσει έξι κριτήρια που αυτά συνεκράτησαν αυτοί που έλαβαν την απόφαση. Ο προφανώς το θέμα της τιμής της έδρας ή του μισθώματος της έδρας δεν ήταν το μόνο κριτήριο. Και νομίζω ότι αν το Συμβούλιο είχε ακολουθήσει αυτό το μοναδικό κριτήριο το προσωπικό ε, στο Λονδίνο δεν θα ήταν ευτυχέ. Δεν μπορεί να εγκαταστήσει κανεί μια υπηρεσία όπω είναι ευρωπαϊκή υπηρεσία σε μια πόλη ή σε μια πόλη σε ένα χωριό, διότι είναι πολύ ακριβό το μίστομα και να μην υπάρχει καμία διασύνδεση με τον κόσμο στον οποίο πρέπει να κινείται η υπηρεσία. Όσον αφορά την συνέργεια μεταξύ των ε, υπηρεσιών, πιστεύω ότι η τροπολογία που προτείνουμε με τον κύριο Μπάλτς είναι σαφέστατη. Ε, δεν θέλουμε να συγχωνεύσουμε τους ρόλους, τα καθήκοντα, θέλουμε να σεβαστούμε την ε, ανεξαρτησία των ε, υπηρεσιών και να επιτρέψουμε όμως και οικονομίες του προπολογισμού που ήταν και βασική μέρημνα του Αντιπρόεδρου βασική ανησυχία. Ευχαριστώ. Θα κοινοποιήσουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και δίνω τον ε, θέση της Προέδρου στην Κέιτ Σουίνμπορν. Γιατί εσάς δεν σας αρέσει να προεδρεύετε, το ξέρω. Yes. Okay. Thank you. Um, Σας ευχαριστώ όλους. Απροσδόκητη καμπή αυτή για μένα. Ο Μάρκος είναι οπότε θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τα καθήκοντά μας. Η γνωμοδότηση που έχουμε μπροστά μας, η γνωμοδότηση για τα τέλη για οχήματα που χρησιμοποιούν κάποιες υποδομές και αφορά διατάξεις για την φορολόγηση οχημάτων. Εδώ και η γνωμοδότηση ΕΚΟΝ, η θα πάρει το λόγο πρώτο και σκιώδης ο καθένας θα έχουν μέχρι ένα τρίλεπτο ο καθένας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που με απαλλάσσεις από την υποχρέωση να πρέπει να δώσω το λόγο στον εαυτό μου εισηγητή. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την αεροβινιέτα, έχουμε δύο τμήματα πρόταση εισαγωγή του συστήματο βινιέτα και το πρόταση σταδιακή μείωση των ελάχιστων κανόνων σε ό,τι αφορά τα οχήματα και ως μέλος της Επιτροπής μου ανέλαβα την Προεδρία επειδή κανεί δεν την ήθελα. Ε, το διευκρινίζω. Αλλά σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα τη οίκων, δεν είναι τα θέματα τη βινιέτα, άρα θα επικεντρωθούμε στα θέματα ε, φορολογία. Και τα θέματα τη βινιέτα ε, νομίζω μπορούμε να τα αφήσουμε στου συναδέλφου ε, από την Επιτροπή Μεταφορών. Το συζητήσαμε με του συνεισήγητε και χαίρομαι που συμφώνησαν με τη γενική προσέγγιση. Πρώτα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τις προδιαγραφές για τα φορτηγά κατά 20% προκειμένου να ε, έχουν μειωθεί σε μηδενικό συντελεστή σε πέντε χρόνια οι φορολογικοί συντελεστές ε, για τα φορτηγά. Θεωρώ ότι αυτό είναι αφελές πρόταση και πολιτικό εσφαλμένο, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές πέντε φορές πέντε φορές θα πρέπει να κάτσουν οι εμπειρογνώμονες να τα κοιτάξουν. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον κανενός. Γι' αυτό λοιπόν πρότεινα να μην γίνουν πέντε σταδιακές αλλαγές, αλλά πέντε χρόνια μετά από την θέση της εφαρμογής, της εφαρμογή ε, του, νομοθεσίας να μετατραπεί ο ελάχιστος συντελεστής από 100% σε 0% γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και σαφής ε, απαλλαγή από το άχθος ε, για τις προλογικές υπηρεσίες και θα χαιρόμουν αν θα μπορούσατε να με υποστηρίξετε. Ευχαριστώ εισηγητά. Σκιώδης των σοσιαλιστών είναι η Περβάνς Περέζ. Δεν τη βλέπω όμως. Σε αυτή την περίπτωση θα δώσω στον εαυτό μου την Προεδρία όπως και ο Μάρκος. Κανείς δεν ήθελε από την ομάδα μου να ασχοληθεί με την γνωμοδότηση, οπότε σε μένα να απόκειται, που με συντονίστηκα να πω ότι το ECR είναι ικανοποιημένο με την έκθεση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μειώσουν το ειδικό τέλος για τα οχήματα αμέσως μετά θέση σε ισχύ της οδηγίας και να μην περιμένουμε μια πενταετία ούτω ώστε να μειώνονται ετησίως ε, κατά 20% τις φορές. Αυτή τέριαζε με μια άλλη πρόταση που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Μεταφορών και δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, εισφορά που καταβάλουν αυτά τα βαριά οχήματα και να καταληφθούν βινιέτε. Θέλουμε να υπάρχει ευελιξία, ώστε να υπάρχει συνεχή εισφορά χρονική, όπω για τα βαρέα οχήματα που επιβάλλεται στον ΕΒ, αλλά συμφωνούμε ότι αν τα χρονικά τέλη θέλουμε τελικά να εξαλειφθούν για ένα τέλη που βασίζονται στην απόσταση, αυτό θα πρέπει να ταιριάξει με μια εξάλληψη με την παρόλο του χρόνου ε, του VED. Λοιπόν, Επιτρέπεται τώρα μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη αμέσως να μειώσουν αυτό το τέλος και να μην επιβάλλουν διπλό φορολογικό άκθο επί των, οχημάτων, των βαριών οχημάτων. Πάμε τώρα στο στον Ραμό Τρεμόζα, εισηγητή του Ισάλντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, ε, κύριε συγητά. Θέλουμε μια στρατηγική για την Ευρώπη που στην κίνηση, σε κίνηση που ξεκίνησε πέρσι. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη στρατηγική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των γερασκόντων δικτύων μεταφορικών. Έχουμε λάβει υπόψη και τη Συμφωνία του Παρισίου το κλίμα. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε γρήγορη μετάβαση προ καθαρή ενέργεια. Ναι, Επίση, για να μειώσουμε την ε, ρήπανση ατμόσφαιρα και θα πρέπει και να μειώσουμε συμφόρηση στι πόλει και στα αυτοκινητοδρόμου. Η οδηγία αντικαθιστά τα βαρέα, τη φορολόγηση βαρέων οχημάτων ε, μέσω διοδίων και τελών χρήση. Αυτή η πρόταση παρουσιάζεται μάλλον μια πρόταση που προωθεί την εφαρμογή των διοδίων. Μια μορφή τελών διαδρομή που βασίζονται με τη ε, διάρκεια του ταξιδιού. συμφωνώ με την αρχή ο χρήστη πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει στην εκλογική μου περιφέρεια και στο κόμμα μου είμαστε υπέρ ε, μια ευρωβινιέτα. Δηλαδή ο χρήστη να, να πληρώνει τι χρησιμοποιίε που χρησιμοποιεί και να χρησιμοποιεί επίση και για τη ρήπανση. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλό ε, εύρυθμο μεταφορικό σύστημα για την ενιαία αγορά. Είναι βασικό όλοι οι χρήστε, ε, οι κάτοικοι και μη κάτοικοι, πρέπει να εργαστούν για μείωση στρεβλώσεω του ανταγωνισμού και να μην υπάρχει διάκριση βάσει εθνικότητα των οδηγών. Επίσης πιστεύω ότι τα χρήματα που παράγονται από τις εισφορές που καταβάλλουν βαρέα χήματα πρέπει να επανεπενδύεται σε υποδομές οδικές και στα σχετικά δίκτυα. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα χρήματα για βελτίωση του δικτύου και να μην χρησιμοποιούνται αλλαχού. Καταλαβαίνω ότι ο εισηγητή θέλει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στη δική εξάλληψη των ελάχιστων ποσών και έτσι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερε μειώσει σε λιγότερα βήματα. Ε, το κατανοώ ότι πρέπει τελικά να βρούμε κάποιο συμβιβασμό όσον αφορά του στόχου και ταχύτητα τη μετάβαση. Ε, δεν είμαι δογματικό για αυτή τη θέση. Πρέπει να έχουμε υπόψη να μιλήσουμε μόνο με το γενικό στόχο τη προτάσεω, δηλαδή να κινηθούμε προ ε, καθαρότερη ενέργεια, πιο δίκαια τέλη για τη χρήση των ε, δρόμων και να βοηθήσουμε να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση και η συμφόρηση στι αυτοκινητόδρομου και πόλη. Ευχαριστώ. Παλώμα Λόπε. Γκουε. Δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της τη Σπαναλόπες να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Είμαστε σίγουροι ότι το έργο, η συνεργασία με του και τους θα μα οδηγήσει σε καρποφόρα αποτελέσματα, ολοκλήρωση των εργασιών. Είναι σημαντικό για μα ε, να είμαστε κοινωνικά δίκαια και να λάβουμε υπόψη και πτυχέ του περιβάλλοντο στην οδηγία και να επιβάλλουμε σχετικά μέτρα. Συμφωνούμε με το γενικό όραμα του εισηγητού, δηλαδή κυρίω συμφωνούμε με την αρχή ο Χρήστη πληρώνει, και την ανάγκη να μειωθεί η συμφόρηση και οι εκπομπές. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη κοινωνικέ και περιφερειακές διαστάσεις. Οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να ε, μειωθούν ούτως ώστε να μην βρίσκονται σε ισχυρή θέση κάποιες χώρες. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθηθούν να λειτουργούν κανονικά ούτως ώστε η χρήση των διοδίων και οι αλλαγέ για την χρήση να μην επηρεάζουν τι μικρέ επιχειρήσει και τι ντόπιε κοινότητε. Αυτή η οδηγία θα μπορούσε να έχει σε διάφορε περιφέρειες στην Ευρώπη πολύ διαφορετικά αποτελέσματα αν δεν δώσουμε προσοχή σε αυτά τα πράγματα όπω είναι οι ιδιαιτερότητε γεωγραφικέ, οι μεταφορικέ υποδομέ, ή οι συγκεκριμένοι στόχοι κάθε προϊόντο. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιλέξουν ταχύτητα και τα βήματα σταδιακή εξαλείψη των τελών βάσει περιφερειακών ιδιαιτερότητων και διοικητικού κόστους. Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην επεκτείνουμε τη χρονική περίοδο που προβλέπετε. Σε κάποια φάση θα πρέπει να ακολουθήσουμε προσεκτικά, παρακολουθήσουμε προσεκτικά τι θα γίνει με τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο που θα συλλέγονται από τα διόδια. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση των πόρων. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση στα κράτη-μέλη πλευρά εισπράξεω και φορολόγηση. Θα πρέπει να ξέρουμε πού πάνε ακριβώ τα έσοδα από τα διόδια. Ο κανονισμό πέρα των γενικών στόχων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε είδου επιχείρηση θα πρέπει να ε, μπορεί ε, να ασκεί τι δραστηριότητέ τη με το σωστό τρόπο. Αυτά θα αντικατοπτρίζονται στι τροπολογίε μα, επειδή είναι πολύ σημαντικό για μα να ε, προωθήσουμε την υποστήριξη των επιχειρήσεων και μια ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει όλου. Θα κάνουμε τις σχετικές τροπολογίες ή τις κοινωνικές προτεραιότητες και συνεργαστούμε στενά με τον εισηγητή όσον αφορά αυτή την γνωμοδότηση της ΑΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους, κυρία Κετό. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Όπως είπε, ε, και εγώ συμφωνώ με ότι πρέπει η ΕΚΟΝ θα πρέπει να γνωμοδοτεί μόνο στις αρμοδιότητες της ΕΚΟΝ για τα θέματα φορολογικά και δεν θα πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο στα θέματα της κινητικότητας από αυτό αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Μεταφορών. Όμως επί του περιεχομένου δεν υποστηρίζουμε την προσέγγιση που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα να καταργήσουμε την ετήσια φορολόγηση των οχημάτων. Για μα η φορολόγηση των οχημάτων δεν θα πρέπει να επικαλύπτει και με τα τέλη που επιβάλλονται βάσει αποστάσεω, θα πρέπει να συμπρωματικό συμπληρωματικό έσοδο και θα δημιουργήσει τα σωστά κίνητρα για να δημιουργήσουμε ε, τι συνθήκε για πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών θα ρηπαίνει λιγότερο και να μειώσουμε και τη συμφόρηση. Ε, τα διόδια που συνδέονται άμεσα με την χρήση των δρόμων, την απόσταση που χρησιμοποιείται, είναι κάτι που μα βοηθά να πετύχουμε του στόχου του πακέτου κινητικότητα. Αυτό δεν αποκλεί όμω τη φορολόγηση όσον αφορά οικονομικέ, περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ συνέπειε του κύκλου ζωή των οχημάτων. Και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όσον αφορά και την οικονομία και όσον αφορά τι δεσμεύσει ανά τη Συμφωνία των Παρισίων. Γι' αυτό θέλουμε πιο βιώσιμη εναρμόνιση και σχετικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο που θα έχει ο κύκλο ζωή των οχημάτων στην οικονομία και σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά όσον αφορά την παραγωγή του και χρήση του, το βάρο και όγκο του οχήματο να λαμβάνεται υπόψη, αντίκτυπο για το κλίμα και κυρίως εκπομπές στο άνθρακα και κατάργηση των κινήτρων όσον αφορά τα εταιρικά οχήματα για την ιδιωτική χρήση. Προτιθέμεθα να υποβάλουμε τροπολογίες σχετικές τροποποίηση των πινάκων που είναι στο παράτημα της εκθέσεως να απορρίψουμε την ιδέα της μειώσης της φορολογίας μέχρι το 2024 στο 0. Ανταυτού θα υποβάλουμε τροπολογίε στην αρμόνιση τη φορολόγηση όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μέχρι να φτάσει αυτή η χρονιά. Θα υποβάλουμε τροπολογίε όσον αφορά τι ιδεολογικέ σκέψει που τα αλλαγέ. Προσβλέπουμε σε κάποιε ενδιαφέρουσε συζητήσει με άλλου και όλου και είμαι σίγουρη θα καταλήξουμε σε καλά συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μόλι. Έχουμε κάτι the eye. Δεν βλέπω, άρα να σας δώσω κάποια στοιχεία για την ε, έκθεση αυτή. Επειδή η αρμοδιότητα αποκλειστική έχει η Επιτροπή Έκονα, ο Πρόεδρος προτείνει στην ε, τράνα να λάβει υπόψη τις τροπολογίες χωρίς να τις ε, τροποποιήσει για όσους ε, συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση. Αυτό έχει νόημα. Η προθεσμία είναι 7 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα και εξέταση των ε, τροπολογιών και ψηφοφορία στην Ήτρε στις 24 Απριλίου προβλέπεται. Και τώρα θα δώσω και πάλι... Α, ναι, θα δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει την εξέταση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους Κιώδης. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε μια απλή λύση ε, συνενετική. Πάντως πιστεύω πως το περιεχόμενο είναι πολύ πιο ε, δίκαιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούμε να το συζητήσουμε στις, ε, στις συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Πάμε στις ψηφοφορίες. Colleagues, may I ask you to take seat and uh, put your voting card into the machine and Θέλετε να βάλετε τις κάρτες σας και να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. No, I need I need this. One EPP e από το ΕΛΚ παρακαλώ. Δύο. Δύο υπεράριθμοι από το ΕΛΚ, συνάδελφοι. πραγματικά μέλη παρακαλώ να μην ψηφίζουν. Κατανοώ ότι συμμετέχετε στην πολιτική ανταγωνισμό. Αλλά πρόεδρε. Πρόεδρε. Δεν έχω την κάρτα μου. Την άφησα στην άλλη αίθουσα ψηφοφορία. Ναι, θα μετρήσουμε την ψήφο σα. Ε, έχουμε δύο άτομα από το EFTD. Δύο ψήφου. Μάλιστα και ένας χωρίς την κάρτα του. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ Σας παρακαλώ, Μπούρκχαρτ, για σου. Ανάλαβε τα καθήκοντά σου. Να ψηφίσουμε. Έκθεση για το ECN Plus. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά, οι σοσιαλιστές παρακαλώ ψηφίζουν. Κατά. Υπέρ. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Μην καθυστερείτε για να βλέπω. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά φαντάζομαι ότι θέλετε έλεγχο. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Βέρνερ, τον πρόεδρο να πιστεύεις. Ήμκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά Έλεγχος για την 116 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 με προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ. Όχι, όχι, σε ισχυρός. Η προφορική τροπολογία λοιπόν απορρίπτεται, γιατί υπάρχει ένσταση. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό χωρίς προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Άποχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά αυτό ελέγξουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Την 219. Πού πήγε η Άλτα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 245. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά Θα πρέπει να ελέγξουμε παρακαλώ τον 250. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 252 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται και ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε παρακαλώ. ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία. 2.53 και 30 της σύμκο Υπέρ. Κατά. Το έλκυν υπέρ. Εγκρίνεται. Η 254 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 84 και η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 27 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Νομίζω ότι εσείς απορρίπτεστε. Κύριε όχι εγώ προσωπικά. 36 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την 108. Πέρασε. Απορρίπτεται με μία ψήφο. 14 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά Απόχε. Το ECR που χάθηκε. Έλεγχο. Ελέγχουμε παρακαλώ. Είναι κατά. Πέρασε. απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα να ψηφίσουμε επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. η ψήφη υπέρ, η ψήφη κατά, μία αποχή. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Μάλλον, όχι, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Έχουμε να ψηφίσουμε και την έναρξη των διαπραγματεύσεων βάσει της έκτασης όπως ανακρίθηκε. Και για τη σύνθεση της ε, ομάδας διαπραγμάτευσης. Τον πρόεδρο, του Σκιώδης και τον εισηγητή. Με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, ψηφίζουμε a rapporteur <laughs> yeah, I said in the wrong order. Mr. others. Το κύριο και λοιπόν. Πέρας. Plus we have to Αλλά έχουμε να προσθέσουμε τον κύριο Κόμπορν. Ψηφίζετε. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. 46 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 3 οι Συγχαρητήρια στον <coughs> εισηγητή και στη διαπραγματευτική ομάδα. Και τώρα να περάσουμε στο σχέδιο έκθεσης για τη συστάση του Συμβουλίου για την διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αρχίζουμε με μια προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε να την παρουσιάσετε. Υπερβάνω Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μόλις αυτές ε, στους συντονιστές είχαμε μια μακρά και σημαντική συνεδρίαση στη συνέχεια της ακρόασης που οδήγησε την ομάδα μου να προτείνει μια συμπλήρωση για το ψήφισμα που εσείς υποβάλλετε ως εισηγητής και που οδηγεί μέσω μιας προφορική ε, τροπολογίας να ζητήσουμε να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία. Θεωρούμε ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες ενεργεί το Συμβούλιο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σέβεται το πνεύμα της συνθήκης, διότι ενώ είχαμε μια ανακρόαση άτυπη, μέσα στην οποία μέσω μιας έκφραση που εσείς χρησιμοποιήσατε αξιολογήσαμε την ποιότητα των δύο υποψηφίων αλλά προφανώς αυτό δεν εισακούστηκε στη συζήτηση στο Συμβουλίο και δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που πρέπει να τηρηθεί, ξέρουμε ότι σημαντικές ε, και διορισμοί θα έρθουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα και θεωρούμε πως αυτή η διαδικασία θα πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να ξεκινήσουμε σχετική συζήτηση με το Συμβούλιο γιατί αυτό καθορίζει και την ψήφο της ομάδας μου. Ευχαριστώ το σύνολο των πολιτικών ομάδων που υποστήριξαν την πρωτοβουλία μας ώστε να τροποποιηθεί προφορικά αυτή η πρόταση. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ανησυχία σε σχέση με την ισορροπία των φύλων, τη διαδικασία επιλογή, τον ε, χρονισμό της, του διορισμού και την πολιτική ανεξαρτησία, απαιτεί ότι το Συμβούλιο να, μπει, να προβεί σε διάλογο με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση τη διαδικασία για του επερχόμενου διορισμού. Αλλά δυστυχώ δεν είχα το χρόνο να συζητήσω με την ομάδα μου επί τη βάση αυτή τη τροπολογία, που βεβαίω μπορεί να οδηγήσει στο να αλλάξουν οι απόψεις ε, ορισμένων. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ε, μια διακοπή κάποιων λεπτών για να μπορέσω να διαβουλευθώ με την ομάδα μου. Σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά. Διάλειμμα. I understand the coordinators, coordinator as the Group wants to make a Λοιπόν, θέλετε να κάνετε μια δήλωση. Ε, πάμε στην πρώτη προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περβάσε σύντομα. ευχαριστήσω το σύνολο των ομάδων για τη στήριξή τους για αυτή την προφορική, αλλά Πρόεδρε ζητώ να δοθεί και σάρκα σε αυτά σε αυτή την, προφορική τροπολογία γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δεσμευτούμε. Δηλαδή η ομάδα μου δεν θα μπορέσει να υπερψηφίσει τον υποψήφιο ούτε καν την αποχή. Θα απορρίψει στην Ολομέλεια την υποψηφιότητα του κ. Τεγκίντο, εάν δεν έχουμε σαφείς μέσα από πλευρά του Συμβουλίου για τη συνέχεια. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ε, μας αγνόησαν εντελώς εμά και το ρόλο μα ως Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να μπείτε σε διαπραγμάτευση με τον κύριο Τάσκη και τον κύριο Σεντενό για τη συνέχεια τη διαδικασία. με συγκεκριμένα αποτελέσματα πριν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, γιατί διαφορετικά θα πρέπει απλώ να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σα ευχαριστώ. Τώρα να ψηφίσουμε τον διορισμό του κυρίου Ντεγκίντο ω πρόεδρο, ως αντιπρόεδρο της ΕΚΤ είναι ε, μυστική η ψηφοφορία, οπότε ψηφίζουμε. Two EPP too many. Δύο παραπανίσχυ ΕΛΚΑ. Okay. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρα, 14 κατά και 13 αποχές. The report is adopted. Of course it's... Εγκρίνεται η έκθεση βέβαια. Όπως βλέπετε οι αποχές είναι πολλές και τα, η ψήφη κατά είναι το ίδιο νούμερο με τους ε, ε συν, με τα υπέρ. Θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια λοιπόν πριν ε, ε, το Μάρτιο βασικά. Συγχαρητήρια και βέβαια επί τη βάση της εντολής αυτού του κειμένου που μας δίνει αυτό το κείμενο θα ξεκινήσουμε συζήτηση με το Συμβούλιο και το Eurogroup για να δούμε πώς θα βελτιωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με την προφορική που μόλις υπερψηφίσαμε, ευχαριστώ και τώρα Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ε, draft opinion by Case Wimborne on this Σχέδιο έκθεσης από την κυρία Swinburne για την απαλλαγή σε σχέση με την ε, ΙΟΠΑ. όχι, πρώτα την ΕΠΑ. ΕΠΑ. Δηλαδή την ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Αρχικό κείμενο, παράγραφη 1, ενα υπέρ κατά αποχές, 24 ε, υπέρ κατά αποχές κρίνεται συμβιβαστική α με προφορική ε, των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 4, 17 ε, υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε ένα παραπανήσιο. Όλοι συγγνώμη, πρέπει να επαναλάβουμε. Έφτασε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ψηφίζουμε 17, τροπολογία 17. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ G, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 48 υπέρ, 1 κατά, 4 αποχές, συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην ε, πιαν ΕΙΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. Συμβαστική Β με προφορική υπέρκατα κατά αποχές εκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Vote is closed ψηφοφορίας. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται. closed. Τέλος ψηφοφορία 49 υπέρ. Μία κατά τέσσερις αποχές. Έσμα τώρα, αρχή κινητών αξιών και αγορών. Εσύ, ε, συμβαστική α, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική β, Σύ ε, ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, και ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφορία. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 49 υπέρ, ένας κατά, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. The meeting is closed. Τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ.